Um, um, Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση. Να έχω την ησυχία σας παρακαλώ. Με χαρά σας καλωσορίζω, έχουμε πολλά θέματα. Και βλέπω και βλέπουμε χαρά τους συναδέλφους εδώ. Καλώς ορίζω και όλους ε, τους θεατές που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Ελπίζω να έχετε δει και το δελτίο το ενημερωτικό που έχουμε δημοσιεύσει. Όποιος το θέλει μπορεί τακτικά από το διαδίκτυο να εγγραφεί και να του το αποστέλουμε. Η, στο, το ιστότοπος της ε, Επιτροπής μας είναι όλο και πιο ενημερωμένος. Έχουμε, χάρη στον κύριο Αρίας που είναι εδώ, ένα ειδικό ιστότοπο ε, που παρακολουθεί την ηλεκτρονική οικονομία με όλα τα θέματα και επίσης θα μας απασχολήσουν και θέματα του τριμερούς διαλόγου. Πάντως στην, ε, στο δελτίο τύπου θα δείτε περιληπτικά ενημέρωση για τα θέματα που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση και τον τριμερή διάλογο. Αυτά ως προς τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Σημερινή και αυριανή. Μια αλλαγή. Γιατί έχουμε βάλει μία ε, ένα σημείο για τη γνωμοδότησή μας για την Επιτροπή, προς την Επιτροπή των Μεταφορών για τις υπηρεσίες εδάφους. Η Επιτροπή των Μεταφορών δεν δείχνει να είναι διατεθειμένη να τροποποιήσει την εκθεσή της, ως εκ τούτου δεν υπάρχει και εμείς λόγος να τροποποιήσουμε τη δική μας νομοδότηση. Άρα θα μείνουν τα πράγματα όπως έχουν και θα σας ενημερώσουμε μετά το πέρας της ψηφοφορίας για τις κλινικές δοκιμές. Ε, συζήτηση για τροπολογίες. Να δω αν έχω τίποτε άλλο. Έχουμε ενημερώσει τα μέλη με ένα σημείωμα για τις ε, παρατηρήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ως προς τον έλεγχο της χρήσης ε, των προϊόντων καπνού. Αυτά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και σε διάφορες γλώσσες για να παρακολουθούμε την, ε, τις εργασίες μας πρακτικά δεν έχουμε να εγκρίνουμε και ως εκ τούτου μπορούμε να πάμε στο πρώτο θέμα. Ενημέρωση για τους ε, τριμερείς διαλόγους που βρίσκονται να εξελίξει. Κυρία Ρόιτοβα, θα ενημερώσω εγώ για τις χθεσινές συζητήσεις, για το νέο, το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Η σειρά που ακολουθούμε είναι η εξής. Πρώτα έχουμε τον τελωνιακό κώδικα ε, που θα παρουσιάσει ο κύριος Φαπ νομίζω. Γιατί Αντικαθίσταται στην αρμόδια συνάδελφο. Έχουμε τις δημόσιες προμήθειες, τις αναθέσεις και θα τοποθετηθώ εγώ για το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Και ξεκινούμε με τον τελωνιακό κώδικα, με τον κύριο Σουάπ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που έχω την ε, ευκαιρία εγώ σήμερα να μιλήσω για τις εξελίξεις του τριμέρου διάλογου για τον τελωνιακό κώδικα. Εάν κάτι έχω λησμονήσει σε σχέση με τα όσα μου έχει αναθέσει η κυρία Ντεγκρή, παρακαλώ να μου το υπενθυμίσετε. Κάνω λοιπόν την παρουσίαση. Η Κωνστός μου έδωσε ένα σημείωμα όπου μου λέει ότι το κύριο θέμα των συζητήσεων για τις 19 Μαρτίου στον τριμερή διάλογο έχει να κάνει με την προσαρμογή στη συνθήκη της Λισαβόνας και, τους, των, και εφαρμοστικών κανόνων για τον ε, τελωνιακό κώδικα, των εκτελεστικών διατάξεων καλύτερα, και έγινε μια ανταλλαγή απόψεων στη συνέχεια για να εξεταστεί το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εναπομείναντα θέματα. Ε, συζητήθηκε επίσης οι, ε, οι κανόνες προελεύσεως και άλλα θέματα και κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, δηλαδή Μόν Μάλκον, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να ε, αφαιθούν και μια τεχνική συνεδρίαση, τεχνικού τύπου συνεδρίαση, πλην του θέματος του προσορισμού της προελεύσεως τα θέματα που δεν έχουν επιληθεί. Μετά τη συνεδρίαση η συγγήτρια ενημερώνει το Συμβούλιο για τα θέματα που θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τον τριμερή διάλογο και κυρίω όσον αφορά τον ε, εναρμονισμένο τελωνιακό κώδικα και ζητεί παράταση της προθεσμίας που είχε οριστεί από την εντολή της ΣΥΜΚΟ στις 21 Φεβρουαρίου. Αυτά έχω να πω, Πρόεδρε. Και με στη θέση σας. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε κύριε Σφάμπ. Και μια που το είπατε, έχω να σας αναφέρω ότι θα έχουμε και στις 10 Απριλίου ακόμη ένα τριμερή διάλογο, οπότε τότε θα δούμε πώς θα δημοφιλονιστικά τα πράγματα και φυσικά ελπίζουμε τελικά να βρεθεί μια λύση, ιδίως όσον αφορά αυτές τις εφαρμοστικές πράξεις και είπαμε αυτά να ζητηθούν οριζόντια μια που ανακύπτουν σε κάθε τριμερή διάλογο. Γιατί πρόκειται για 20 όρους και προϋποθέσεις που αφορούν αυτές τις πράξεις. Και άρα είναι κάτι το οποίο αναφέρεται στο βασικό κείμενο της οδηγίας. Σας ευχαριστούμε, εν πάση περιπτώσει. Έχει κάποιος κάποια ερώτηση. Sessions, uh, and I give the floor to Philippe Jouvin, our rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Bien, là aussi... Euh, Monsieur Jouvin. Σα υπενθυμίζω ότι ε, και προκειμένου έχουμε θέμα του τριμερού διαλόγου και εσείς συμμετέχετε και ως σκιώδης συζητητής λάβετε υπόψη αυτά που έχω να σας πω Οπότε έχουμε αυτή την εντολή για τη διαπραγμάτευση. Έχουν προγραμματίσει τέτοιε τέτοιες επαφέ. επαφές. Πρώτα-πρώτα είναι η έκθεση Ταραμπέλα, 12 Μαρτίου στο Στρασβούργο. Και έχουμε τρει τεχνικέ συναντήσει με το Συμβούλιο και προβλέπεται για αυτή την εβδομάδα στι 20 Μαρτίου ακόμα μια τέταρτη συνάντηση έχουμε προτείνει συμβαστική λύση στο Συμβούλιο όσον αφορά τις γενικές αρχές οπότε τουλάχιστον για τις τεχνικές συναντήσεις τα πράγματα πάνε καλά και θα πρέπει να ε, θεωρήσουμε ότι είναι πάρα πολύ θετικά ε, τα όσα έχουν εισφέρει οι σχεδόν και τα κείμενα όλων των πλευρών τελικά ήρθαν να συμφωνήσουν. Στις 12 Μαρτίου είπαμε ποιο είναι ο ορισμός της παραχώρησης, ιδίως όσον αφορά την χρήση αυτών των, δύο, των τριών λέξεων που ε, συζητούμε. Πρώτο πρώτο procurement, δεύτερον acquisition και η λέξη consent Οπότε έχουμε ε, συζήτηση για τον ορισμό του οικονομικού κινδύνου, της διαφάνειας Οπότε τώρα τελικά θα ξεπεραστούν φαντάζομαι οι δισταγμοί του Συμβουλίου σχέση με τις δικές μας προτάσεις. Επίσης συζητούμε και για το κατόφλι, κάτι που είναι πιο δύσκολο γιατί έχουμε αυτά τα 8 εκατομμύρια ως κατόφλι, το οποίο από κοινό καθορίστηκε. Από ό,τι φαίνεται έρχεται σε αντίθεση με κάποιες διεθνείς συμφωνίες και επομένω θα πρέπει να συζητηθεί όπως και τα αποκλειστικά δικαιώματα που τα συζητούμε με το Συμβούλιο, οπότε και είναι προκειμένο ε, νομίζω ότι θα βρεθεί μια, ε, μια λύση συμβαστική. Τώρα όσον αφορά την διάρκεια της παραχώρησης είναι πολύ βασικό θέμα και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός στο κείμενο. Επίσης, ε, στάλει μια πρόταση συμβασμού χθε στους σκιώδους ηγητές. Έστειλα φωτογραφία μου για, όσον αφορά τα κατόφλι ή το κατόφλι εκεί που συνεχίζεται αυτή η το κατοφλι εκει που συνεχιζεται αυτη η προσθετή με το Συμβούλιο για τον λόγο που σας είπα, και οπότε γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι διαπραγματεύσει πάνε καλά και ε, διαπραγματευόμαστε στα προβληματικά σημεία ένα συμβασμό. Επίσης να δούμε τι, πώς θα εμβαθύνουμε σε κάποια σημεία. Δηλαδή θέλουμε εμείς να υπάρχει ένα κειμένο ρεαλιστικό, σαφές, κατανοητό και έτσι θέλουμε να συμβάλλουμε ως κοινοβούλιο σε αυτό το νέο νομοθέτημα. Αυτά όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Good. Thank you very much uh, for that. Um, anybody got... Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Έχει κάποιες ερωτήσεις προς τον κύριο Ζουβέν όσον αφορά την πρόοδο των επαφών για τις παραχωρήσεις. Πάμε τώρα στην έκθεση Ταραμπέλα για τους διαγωνισμούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. 6 Μαρτίου έγινε ο πρώτος τριμερής διάλογος σε καλό κλίμα. Όλοι φαίνεται ε, να δείχνουν ε, κατανόηση προς τους άλλους ε, και χαιρετίζω και την προσπάθεια προσέγγισης της Κομισιόν εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερες διαφορές. Όμως διαπιστώνω ότι το Συμβούλιο παραμένει ε, στις ε, θέσεις του ε, και δεν είναι έτοιμο να κάνει κινήσεις έτσι ώστε να προσεγγίσει το κοινοβούλιο. Το λέω, το είχα πει και από πριν γιατί ήταν η εντύπωσή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει το είδα και μετά από τις συναντήσεις. Πάντως είχαμε και εκεί κάποιες πρόοδους, είχαμε τη δυνατότητα να επιμείνουμε ότι στο μέλλον και μέσω των τεχνικών ε, συναντήσεων ε, να βρούμε έναν καλό ρυθμό ε, θα φτάσουμε μέχρι τον Ιούνιο, ελπίζω να μην ξεπεράσουμε και τον Ιούνιο, ε, και ε, νομίζω ότι καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι όταν φτάνουμε στον τριμερή διάλογο έτσι ώστε να ξέρουμε αμέσως ποια είναι τα σημεία στα οποία μπορεί να υπάρχει εμπλοκή και πώς μπορούμε να, τελειώ... να προχωρήσουμε. Ε, στον πρώτο τριμερή διάλογο είχαμε συζήτηση για το κλάστερ 1 όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας δηλαδή συζητήθηκε το θέμα των διαπραγματεύσεων, το ηλεκτρονικό ε, διαβατήριο. Ίσως το είδατε διαβάζοντας το κείμενο που ενέκρινε το Συμβούλιο ε, ότι η προσέγγιση του Κοινοβουλίου δεν είναι τόσο ολοκληρωμένη όσο του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο θέλει πραγματική ενιαία αγορά με πλατφόρμες ε, οι οποίες ε, θα είναι διασυνδεδεμένες και βέβαια η δυσκολία εκεί είναι μεγαλύτερη. Εδώ έχουμε 7 πολιτικές ε, ομάδες, και έχουν 27 χώρες οι οποίες ενδεχομένως η καθεμία περιχαράσει τη θέση της περισσότερο από ότι εδώ οι πολιτικές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει αυτή η ηλεκτρονική ε, διαδικασία εάν, ε, ε, εάν θα εφαρμοστεί μονάχα μερικώς θα κατακαιρματίσει την αγορά και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε. Πολύ συζήτηση γίνεται, προσπαθούμε να βρούμε βεβαίω συμβαστικέ λύσεις. Τώρα η υποχρεωτική εφαρμογή όλων των διαδικασιών ε, ε, βεβαίως θα πρέπει να είναι διαφανής ε, και ε, οι υποχρεωτικές αυτές οι διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων ε, οι εξαιρέσεις που ζητάει το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι σαφείς, θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ε, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί η ρήτρα της εμπιστευτικότητας ε, σαν πρόσκομα. Το ηλεκτρονικό διαβατήριο αυτό θα πρέπει να, είναι, να χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορεί να υπάρχει διαλειτουργικότητα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όλες τις πλατφόρμες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κιώδης ε, για την ε, στήριξη ε, επόμενη τριμερής ε, συνάντηση είναι στις 26 Μαρτίου. Εκεί θα είναι πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Θα συζητήσουμε το κλάστερ 5, ε, καλύτερη ε, δυνατή συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το άλλο κλάστερ είναι το κλάστερ 2, στρατηγική σημασία των δημοσίων προμηθειών. Αυτά μπορώ να σας πω κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. καλά κάνετε και αναφέρεστε και στη γενικότερη δυναμική των συζητήσεων, ε, γιατί πραγματικά και η τεχνική προετοιμασία είναι πάρα πολύ μεγάλη και η τεχνική εργασία που γίνεται πριν είναι πολύ μεγάλη. Απ' την άλλη πλευρά είναι πολλές οι χώρες, είναι δύσκολο ε, να βρεθεί ε, έτσι άμεσα μια κοινή θέση και βεβαίως και το Κοινοβούλιο δεν αφήνει να περάσει τίποτε, όλα τα συζητάει. Βλέπω ότι είναι η κυρία Ροϊτόβα ε, μαζί μας. Μπορεί να μας μιλήσει για το νομοθετικό πλαίσιο. Να μας ε, κάνει μία σύντομη παρουσίαση, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Κυρία Ροϊτόβα, θέλετε να μας ε, πείτε δύο λόγια για τον τριμερή διάλογο που είχατε χθες το βράδυ και το νέο πακέτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης και τον Πρόεδρο Χάρμπορ γιατί ε, νομίζω ότι χθες ε, καταφέραμε να κάνουμε κάτι ανέλπιστο. Ε, δηλαδή να προσεγγίσουμε κατά 99% το κλείσιμο της συζήτησης για μια οδηγία κλειδί που αφορά το Good Package του 2008. οι τεχνικές συζητήσεις στέφθηκαν από επιτυχία ε, και όλα όσα ψηφίσαμε εδώ τελικά ε, βρήκαν τη θέση τους ε, στην τεχνική, στις τεχνικές συναντήσεις και βεβαίως για να μην μιλήσω εδώ, να μην μακρηγορήσω θα σας ετοιμάσω έτσι ένα γραπτό κείμενο Το Συμβούλιο επιθυμεί ε, οι ομάδες εργασίας που υφίστανται αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της επιτροπολογίας ε, να διατηρηθούν και να ασχοληθούν και με την υλοποίηση κάποιων επιμέρους ζητημάτων του κανονισμού. Όμως ε, δεν είναι δυνατόν να βάλει το Συμβούλιο αυτές ε, τις ε, αρχές να τις υλοποιήσει και να τις βάλει στις οδηγίες γιατί υπάρχει αντίβαση προς τις, αντίφαση με τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Λισαβόνας και με το πρωτογενές δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να πούμε ότι στις συζητήσεις ε, έχουν ε, προσκληθεί και εθνικοί εμπειρογνώμονες ε, και γίνεται διαβούλευση μαζί τους για την υλοποίηση και εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Πάντως είναι πολύ θετική και επικοδομητική η στάση όλων. Εάν ε, οι αποφάσεις της επόμενης Παρασκευής ε, ταυτίζονται με τα όσα αποφασίσαμε εμείς, ε, μπορούμε να εγκρίνουμε το κείμενο έτσι ώστε τον μήνα Μάιο να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια και θα έχουμε μπροστά μας αυτό το 5% σε σχέση με τις 8 οδηγίες που ακόμα παραμένουν ε, για τα υπόλοιπα σας είπα οριζόντια και τομεακά έχουμε ε, κλείσει 95%, 95% όχι 99, 95% αυτό το 5% που μένει ε, θα νομίζω ότι έχουμε δυνατότητα να το καλύψουμε. Όσον αφορά τώρα το υπόλοιπο του πακέτου μπορούμε να το ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. thank you very much. Ευχαριστώ πολύ είχαμε για τα υπόλοιπα τεχνικά ζητήματα μια συμφωνία, γιατί ο υφισταμένος κανονισμό εκπνέει τον Ιούλιο, αλλά έχουμε βρει κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Ε, κάτι άλλο? Καλώ λοιπόν, για να κλείσει το θέμα αυτό, για να είμαστε πλήρε, θέλω να σας πω ότι ο πρώτος τριμερής διάλογος για τα επαγγελματικά προσόντα λαμβάνει χώρα σήμερα. Κυρία Δεγνιό είναι η συγγήτριά μας και έκθεση θα έχουμε στην προσεχή συνεδρίαση. Και στο δικό μου το θέμα θα ξαναρχίσει μάλλον αρχάς Μαρτίου ο τριμερής διάλογος. για τα σκάφη ένας ψυχής. Ελπίζω λοιπόν να δούμε κάτι καλό και από αυτές τις πραγματεύσεις. Κλείνουμε το θέμα αυτό. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο και σημαντικό. Μια νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής μας. Πιστεύουμε ότι είναι καλό να εμπλέκονται οι πάντες τακτικά, να παρακολουθούν τις εργασίες μας. Πολλοί από εσά βέβαια και ως και ηγητές ε, ήδη έχετε ε, την ευκαιρία να παρακολουθείτε ενεργά τα θέματα αυτά. Τώρα έχουμε μια γνωμοδότηση που πρόκειται να ψηφίσουμε αύριο για τις κλινικές δοκιμές, τη σχετική οδηγία, όπου θα παρουσιάσει συμβιβαστικές τροπολογίες μόνο ο εισηγητής. Θα σας παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι και παρακαλώ τώρα τον κύριο στις δικές σας παρατηρήσεις και σχόλια και παρακαλώ τώρα τον κύριο Πουζόη να λάβει το λόγο για τις συμβαστικές του τροπολογίες με την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα και ότι θα, θα τις εγκρίνουμε. Ο κύριος Μπουσόη, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα χρειαστώ πάνω από πέντε λεπτά. Θα είμαστε δυνατόν πιο σύντομος. Είχα πολύ καλή συνεργασία με τους κοιόδης ηγητές, με τους λοιπούς ε, ε, συναδέλφους, με τη γραμματεία. Είναι σημαντικό το θέμα της οδηγίας αυτής, δηλαδή θέλουμε να έχουμε πιο καινοτόμες ε, κλινικές δοκιμές, θέλουμε υποστήριξη για τον ιατρικό κόσμο. Έχουμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες λοιπόν και προφορικές επίσης που ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να μετατραπούν σε, θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές ως ε, συμβαστικές στην πραγματικότητα, αλλά για λόγους τεχνικούς τις καταθέτουμε ως προφορικές. Λοιπόν, σχετικά με το τι μπορεί να είναι ο ορισμός και η κοινοποίηση. Έχουμε διαγράψει το κομμάτι που αφορά τα άρθρα 8, 14, 19, 20 και 23 διότι δεν εξαρτάται από το χρονικό διάστημα, αλλά από το περιεχόμενο ορισμός. Επίσης, συμβασμό έχουμε ως προς τις διαδικασίες και ιδιαίτερα την, τον προσδιορισμό του κράτους ενημέρωσης, reporting member States ενώ υπήρχε μια πρόταση να δοθεί δυνατότητα στα κράτη-μέλη να κρίνουν. Εγώ δεν έχω αντίρρηση σε αυτό, εφόσον όμως στηρούνται τα σχετικά χρονοδιάγραμμα, τα χρονοδιάγραμματα, αυτό προτείνει η Επιτροπή δηλαδή. Και έτσι λέμε ε, να προτείνει ο χορηγός το κράτος μέλος ενημέρωσης, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό και μπορεί το εν λόγω κράτος μέλος μέσα σε τρεις ημέρες ε, να προτείνει ένα άλλο κράτος μέλος. Εάν ε, όχι, θα είναι αυτό που έχει προτείνει ο χορηγός. Επίσης έχουμε την τήρηση πιο αυστηρών ε, εθνικών διατάξεων για με στόχο την προστασία του ενδιαφερομένου και δύο όταν πρόκειται για πιο ευάλωτους, ε, ευάλωτα υποκείμενα. Εδώ δεν έχουμε ορισμό του ποιος είναι το ευάλωτο υποκείμενο. Μετά έχουμε την δεοντολογική προσέγγιση και αξιολόγηση που αφορά τροπολογίες σε διάφορα σημεία του κειμένου και έτσι προσπαθώ με το άρθρο 7α να συνενώσω και το θέμα της ε, αδειοδότησης της δοκιμής και της περαιτέρω τροποποίησης της. Δηλαδή με το συμβασμό ξεκινά η κλινική δοκιμή μόνο όταν έχει η αρμόδια αρχή ε, ξεκινήσει και χορηγήσει την διοντολογική ε, αξιολόγηση ή αδειοδότηση και έτσι μόνο, όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, επισημαίνουμε ότι θα πρέπει αυτή η εδοντολογική ε, αξιολόγηση να καθυστερεί την όλη διαδικασία της κλινικής δοκιμής. Επίσης, όταν μία αίτηση επανυποβάλλεται, ύστερα από μία πρώτη απόρριψη ή απόσυρση, θα πρέπει και αυτή να δηλώνεται, η αρχική δηλαδή απόρριψη ή απόσυρση, αλλά και οι λόγοι της επανυποβολής. Στο 6, συμβαστική τροπολογία 6, ε, προτείνεται περισσότερη ευελιξία σε περίπτωση ε, έκτακτης ανάγκης, με τον ελάχιστο κίνδυνο που προσδιορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, έτσι ώστε να μπορεί να ξεκινήσει χωρίς την ρητή συνένεση η κλινική δοκιμή εφόσον υπάρχει κίνδυνο ζωής. Και βάζουμε την διατύπωση ότι πρέπει η συμμετοχή στις κλινικές δοκιμές ε, να προσφέρει πλεονέκτημα όφελος ανάλογο με τον κίνδυνο ε, ή πάντως μικρότερο από τον κίνδυνο που ενδέχεται να διατρέξει το υποκείμενο της δοκιμής. Συνεχίζω με τροπολογία που υποστηρίζουν οι ε, ομάδες σε σχέση με την αξιολόγηση, με την περίοδο αξιολόγησης την οποία από ένα έτος στην αρχική πρόταση την έχουμε μεταφέρει στα δύο έτη, ώστε να υπάρχει δυνατότητα και για την δημοσίευση σε ένα σημαντικό ιατρικό περιοδικό που χρειάζεται ενδεχομένω περισσότερο χρόνο για τους ε, πανεπιστημιακούς και ερευνητές, ώστε να τους δίνουμε την ευκαιρία να δουν τη δημοσίευση του άρθρου τους σε κάποιο σημαντικό περιοδικό. Στη συνέχεια... Ε, έχουμε την πρόταση του, άρχου, του άρθρου 202, της δικής μου τροπολογίας 202, όπου έχουμε όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν, όλα τα στοιχεία που πρέπει να κοινοποιούνται, που θα πρέπει να επιτρέπουν στους ερευνητές να επαληθεύουν. Για δε τις εμπορικές χρήσεις, όχι δηλαδή την ε, επιστημονική αξιολόγηση, ε, παρουσίαση, 30 μέρες από την δημοσίευση ή από την διακοπή της, ε, από τη δημοσίευση της αδειοδότησης, από την αδειοδότηση, ε, θα πρέπει να είναι το όριο ε, για την εμπορική χρήση. Πάντως θα περιλάβω και στον ορισμό των συμπληρωματικών ιατρικών στοιχείων και προτάσεις σχετικές με αυτές τις τροπολογίες της κυρίας Μακλάρκιν και προτάσεις σε σχέση με την αξιολόγηση των ικανοτήτων των αρμοδίων για την αδειοδότηση και για την ε, υποχρέωση κοινοποίηση όταν γίνεται πολυκρατική ή διεθνική μία κλινική ε, δοκιμή αντί για εθνική και επίσης προτάσεις σχετικέ με τους ορισμούς μπορεί να αποκλίνουν από το ένα κράτο μέλος στο άλλο. Τα έχετε όλα αυτά τα θέματα στους, ε, στα εγγραφά σα. Αυτά είναι λίγο πολύ όσοι έχουμε συμφωνήσει, βελτιώνουν το κείμενο και ελπίζω ότι αύριο στις 10.30 που έχουμε την ψηφοφορία θα μπορέσετε να με υποστηρίξετε όλοι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ισχυρός. τώρα. Κύριε Μακλάκιν και κύριε Ρούλα, εάν έχουν κάποια σχόλια μπορούν να τα υποβάλουν όσον αφορά τις τροπολογίες. Και επίσης να επιβεβαιώσουν το αν συμφωνούν ή όχι με όλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, λέει κύριε Σαλντεμάς, ευχαριστούμε συγκεκριτά για την αναζήτηση λύσεων. Δεν συμβρούμε με όλες τις τροπολογίες. Έχουμε κάποιες προτάσεις. Θα σας τα πούμε αργότερα αφού συνδυάσει η ομάδα εργασίων. Εν πάση περιπτώσει όμως, σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε. Α, συγγνώμη κύριε Ζουβά, πρέπει να δώσω λόγο νωρίτερα. Πρώτα πρώτα πρόεδρε, συμφωνούμε με όλες τις συνεργασίες ε, του Πολυσκηρίου Μπουσόη ε, δεύτερον, υπενθυμίζουμε ότι έχουμε πέντε συμβαστικέ οι οποίε έγιναν προφορικές τροπολογίες ε, για το ζήτησε η γραμματεία της ε, ΙΜΚΟ και θεωρώ ότι κανεί δεν έχει αντίρρηση. Με αυτή, τη μετατροπή δεν λοιπόν να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά. Αλλά δεν υπάρχει αντίρρηση για αυτή τη διαδικαστική μετατροπή. Επίση όσον αφορά τη συμβαστική παριθμών 7 μια διευκρίνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι λέει πρώτα πρώτα ότι η δημοσίευση είναι υποχρεωτική, κάτι το οποίο σήμερα δεν ισχύει. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δημοσίευση που να είναι κατάλληλη για το κοινό και επίσης να είναι κάτι κατάλληλο, δόκιμο για τους επιστήμονες οι οποίοι να μπορούν να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα. Όμως, ε, βασικό στοιχείο αυτής της τοποθέτηση, κύριε Μπουσόη, ότι είναι ε, όχι σε, για δύο χρόνια υποχρεωτική αυτή η δημοσίευση γιατί όταν γίνεται κάποια τέτοια εργασία, κάποια δοκιμή, αυτό δημοσίευσε σήμερα στο περιοδικό και μετά υπάρχει μια δημοσίευση πριν ε, στο, στο, στο website, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να, να πάρει κάποιος την ιδέα. Οπότε Γι' αυτό και έχει σημασία το ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η αναμονή. Γιατί υπάρχουν κάποιες μελέτες που δεν είναι το ίδιο σοβαρές. Δημοσιεύονται, αλλά δεν υπάρχει αναγκαία ενημέρωση. Ενώ τώρα, με αυτή την αναμονή, είναι βέβαιο ότι έχει εγκριθεί από την προσωπική κοινότητα. Οπότε έτσι, με, με αυτόν τον τρόπο τώρα, θα είναι πιο κατανοητή κατάσταση στον κόσμο, στο κοινό. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Κυρία Ρούλη. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία, για την πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Μπούσο και φυσικά δεν θα ε, αντιδράσουμε στην υποβολή των προφορικών τροπολογιών. Δεν έχουμε αντίρρηση. Ε, για τι συμβαστικέ τροπολογίε πάντω, κάποιε από αυτέ θα υποστηρίξουμε και έχουμε κάποιε επιφυλάξει όσον αφορά την ψηφοφορία. Θα γνωρίζετε ασφαλώ ότι πιστεύουμε ότι χρειάζεται να διατίθενται πολύ περισσότερε πληροφορίε στην κοινή γνώμη, χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Σε αυτό είναι οι επιφυλάξει μα και ανάλογα με το ε, πώ θα προκύψει, προκύψουν και οι θέσει μα με του συναδέλφου μα που βρίσκονται στην Επιτροπή του Περιβάλλοντο, θα προσδορίσουμε και τι θέσει μα για τι ε, ψηφοφορίε. Ναι, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η εργασία μας για το θέμα αυτό και ευχαριστούμε τον εισηγητή για την συνεργασία του. Έχουμε όλες αυτές τις σημαντικές τροπολογίες και ελπίζουμε η κατάσταση να βελτιωθεί. Έχω μια προφορική τροπολογία για τον ορισμό του άρθρου 2. Επίσης, για την Ανεξάρτητη Επιτροπή Διοντολογίας. Ε, πάρα πολύ καλό το συμφωνήσαμε και για το άρθρο 5. Τώρα τα πράγματα έχουν ξεκαθαριστεί. Όσον αφορά τις κοινοποιήσεις, επίσης συμβαστική 7. Επ' αυτής εκεί έχουμε την απαλυφή ενός εδαφίου που είχε στην αρχή πρώτα από την Επιτροπή και έτσι τώρα θα έχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις περισσότερη ευελιξία. Πάντως, εγώ θα ψηφίσω υπέρ της τροπολογίας γιατί βελτιώνει το αρχικό κείμενο. Έχω βέβαια και κάποια επιφύλαξη. Πάντως, συνάδελφε, παρακαλώ να ψηφίσετε υπέρ της δικής μου τροπολογίας που αφορά την συμβαστική 6 γιατί έτσι νομίζω ότι για τις δοκιμές μπορούμε να σταθμίζουμε καλύτερα τα υπέρ και τα κατά τους κινδύνους και ελπίζω λοιπόν να παρακαλά καλά για αυτό το ενδιαφέρον αλλά δύσκολο θέμα. Εμεί σα ευχαριστούμε. Κυρία Γκέπχαρτ τη ζητήσει το λόγο. Και επίση όποιο άλλο θέλει μπορεί να σχολιάσει. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συνεργασία. Έχω μια συμπληρωματική ερώτηση για τον κύριο Μπουσόη. Με τη συμβαστική 4 για το 7α καινούριο άρθρο Εκεί λέγεται ότι η αδειοδότηση μιας δοκιμής μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν της εγκρίσεως της αρμόδιας επιτροπής δεοντολογίας. Εγώ είμαι υπέρ της ε, παρέμβαση Επιτροπή Δεοντολογίας, δηλαδή να στείτε η γνώμη της προκαταβολικά. Αλλά εδώ μιλούμε για Εθνικές Επιτροπές Δεοντολογίας. Υπάρχει ορισμός αυτών των επιτροπών. Πρώτον. Δεύτερον, διαθέτει κάθε κράτος μέλος Επιτροπή Διοντολογίας. Και τρίτον, εάν όχι, τότε, και είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι πρόκειται για κανονισμό αυτό θα συνεπαγόταν αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των δοκιμών γιατί, ή όχι, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με θέματα δημόσιας έχουμε να κάνουμε θέματα υγείας των πολιτών μας και δεν θέλουμε να ανοίξουμε θύρες και παράθυρα σε ένα forum shopping, δηλαδή στην δυνατότητα ο καθένας να ε, ψάχνει να βρει τις πιο ωφέλιμες λύσεις, δηλαδή τις λιγότερο δεσμευτικές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος είναι εδώ από την Γενική Διεύθυνση ε, Δημόσιας Υγείας. Εάν θέλετε να λάβετε το λόγο, να μας δώσετε τις θέσεις σας για να προχωρήσουμε σχετικά σύντομα όμως. Και στο συγγνώμη που σας πιέζω, αλλά έχει τελειώσει, έχουμε ξατλήσει το χρόνο μας. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή για την ε, πολύ καλή εργασία του. Παρ' όλα αυτά να υπογραμμίσω δύο σημεία τα οποία είναι σημαντικά για την πρόταση. Πρώτον, ε, πρώτο σημείο σχετικά με την εμπλοκή της ε, Επιτροπής όσον αφορά την αδειοδότηση και δεύτερον τα στάνταρ, τα πρότυπα προστασίας. Ε, για το πρώτο σημείο πρέπει να σας πω ότι υπάρχει η οδηγία πλαίσιο η οποία καθορίζει συγκεκριμένα ε, στοιχεία. Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν για να αποσαφηνίσω ότι η Επιτροπή δεν θέλει, ε, ε, δεν θέλει μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ε, να διασφαλίσει ε, την καλή λειτουργία αυτών των υποεπιτροπών γιατί ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μας να τις ε, διαλύσουμε. από την άλλη πλευρά θέλουμε να χτίσουμε ένα καλό σύστημα διοδότησης σεβόμενη και την, τις παραδοσιακές γνώσεις, της, την τεχνογνωσία αλλά και τις παραδόσεις που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Θέλουμε όλα αυτά να τα ε, ε, καλωσορίσουμε και να τα λάβουμε υπόψη μας όλες ε, οι διαδικασίες όσον αφορά την αδειοδότηση αναφέρονται στο ίδιο το σώμα της οδηγίας. Δεύτερον, η προστασία και τα συνήθη μέτρα για προστασία πρέπει να σας πω ότι μας ενδιαφέρει ο υψηλός βαθμός προστασίας ε, όλων των συμμετεχόντων στις ε, κλινικές ε, δοκιμές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει σαφήνεια κανονισμών. Γι' αυτό ακριβώς εμείς επιλέξαμε το μέσο του κανονισμού. Θέλουμε να είναι ίδια τα κριτήρια κατά την αξιολόγηση των κλινικών δοκιμών, γιατί εάν τα κριτήρια διαφέρουν, τότε η αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι ε, σωστή. Και να σας πω βεβαίως ότι η Κομισιόν με πολύ μεγάλη προσοχή άκουσε την προσέγγιση όλων ε, εμείς. Πρέπει να σας πω ότι στο νέο κείμενο ακολουθούμε ε, στην ουσία το παλαιό κείμενο και οι πρόνοιες ε, δεν έχουν αλλάξει τα υφιστάμενα κριτήρια τα οποία είχε αναφέρει ο νομοθέτης ήδη το 2001 και μη λησμονούμε ότι αυτά τα στοιχεία βεβαίως έχουν προκύψει και από τα υφιστάμενα σε άλλα διεθνή ε, κείμενα. Φυσικά ε, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ο νομοθέτης θέλει όμως να έχει μία ενιαία ε, δέσμοι ε, μέτρων και κανόνων ε, που θα εφαρμόζονται σε όλες τις αξιολογήσεις των δοκιμών. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θέλουν να υπάρξει επικαιροποίηση της οδηγίας για τις κλινικές δοκιμές και ο ακαδημαϊκός κόσμος και ο ιατρικός και επομένως ευελπιστούμε ότι θα οδηγηθεί σε σωστό δρόμο η συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Μπουζόη, ζητώ συγγνώμη που σας δώσαμε τόσο λίγο χρόνο, αλλά δυστυχώς έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Ο κύριος Μπουζόη, δεν θα ολοκληρώσω, απλώς ε, θα απαντήσω στο σημαντικό ερώτημα της κυρίας Γκέπχαρτ. Και επίσης Είμαστε βέβαιοι ότι οι ιδεοντολογικέ αυτές επιτροπέ, ε, οι οποίες, δεν το γεγονό μάλλον ότι δεν περιλαμβάνονται ε, δεν είναι απόρρια του γεγονότος ότι δεν τι θέλει η Κομισιόν. Απλώ εμεί θέλουμε να είναι σαφέ ε, ότι η ηθική αξιολόγηση, η ιδεοντολογική αξιολόγηση είναι εξίσου σημαντική με τι άλλε αξιολογήσει. Μη λησμονούμε επίσης το θέμα τη επικουρικότητα, δηλαδή η κάθε χώρα μπορεί να οργανώσει τη δικιά της ε, διαδικασία εάν ε, ε, σέβεται τα περιλαμβανόμενα και τα χρονοδιαγράμματα της οδηγίας. Δηλαδή μπορεί να γίνει σε ε, επίπεδο περιφέρειας ή επίπεδο εθνικό. Υπάρχει και μια χώρα μέλος ε, η οποία οργανώνει αυτές τις διοντολογικές επιτροπές σε επίπεδο πόλης. Ε, να υπάρχουν λοιπόν αυτές οι επιτροπές αρκεί να σέβονται το γενικότερο πλαίσιο της οδηγίας. Πάρα πολύ ωραία. Θα ψηφίσουμε στις 10 αύριο για το θέμα αυτό και θα δούμε πώς, αν θα περάσουν και πόσες τροπολογίες θα περάσουν. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. να ξεκινήσουμε τη σκέψη ε, για την ε, έκθεση Fox, διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στην εσωτερική αγορά θα ακούσουμε την άποψη κάποιων εμπειρογνωμόνων σήμερα το πρωί, αλλά πάντως πρέπει να τελειώσουμε μέχρι τις 10.30, γιατί έχουμε κι άλλη μία ακρόαση και μόνο μου ότι αυτό εδώ είναι το ξεκίνημα, το άνοιγμα της συζήτησης. Ε, θα έχουμε την δυνατότητα να αξιολογήσουμε την έκθεση Fox. Ε, θα δώσω λοιπόν πρώτα τον λόγο στον κύριο Fox ε, να μας κάνει την πρώτη εισαγωγή. Μετά θα έχουμε την κυρία Πιέτη Κάνεν Ξέρω ότι ενδιαφέρεται πολύ για το θέμα αυτό, άλλωστε έχουμε και φιλανδική αντιπροσωπεία, έχουμε τον κύριο Πικάτο. Um, uh, who I welcome. And uh, then we have Mrs. Schaldemoser, Mr. Kreutzmann, Mrs. Ruler, and Mr. de Jong uh, for all the shadows are here as well. Um, so without more ado, I'm going to give the floor to our rapporteur. Θα δώσω αμέσως το λόγο Ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Um... ευχαριστώ. Can I extend a particularly warm welcome to Mr. καλωσορίσουμε τον κύριο Γκάντο που είναι ο υπουργό που θα μα συγκρίνει από το Γιβραλτάρ. Είναι πάρα πολύ, είναι τιμή μα που εκπροσωπεί στο πρόσωπό του η χώρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επομένω ε, μεγάλη μου χαρά σήμερα ε, σα παρουσιάζω την έκθεση αφού έχω συνενεθεί με όλου του ε, εμπλεκομένου. Ε, από όλου αυτού του ειδικού, στον εθισμό, στα τυχερά παιχνίδια, ε, Και οπότε έγινε μια πρώτη αναλογία ε, απόψεων. Θα προσπαθήσω να καλύψω τόσα άκουσα. Ε, ήταν προσπαθώ να δεν όλα όσα μου είπαν σε αυτό το πρώτο σχέδιο Ξέρετε ότι μα επιτρέπουν οι μόνοι των συντακτών μόνο 6.000 χαρακτήρε όταν έχουμε το πρώτο σχεδό κειμένο και γι' αυτό και δεν επισερχόμαστε σε λεπτομέρειε πολλέ φορέ σε διάφορα ζητήματα για τα οποία μιλήσαμε. Αλλά νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα των τροπολογιών αυτό το, το, το, το πρόβλημα μπορούμε να το λύσουμε. Πάντω η αίσθηση που έχω από την τελευταία ανταλλαγή απόψεων είναι ότι έχουμε από όλε τι πολιτικέ εταιρείε του Κοινοβουλίου διακομματική υποστήριξη σε σχέση με την ε, προστασία των καταναλωτών και πολλοί συνάδελφοι είπαν πάρα πολλά εύστοχα γιατί κάποια κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να προσθέσουν του καταναλωτέ ή περιορισμού που σε, σε, σε, σχέση με τα, με τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Και βέβαια, αν έχουμε κάποιο είδου απαγόρευση ή αν τέλο πάντων έχουμε ε, ε, ε, ένα καθεστώς το οποίο δεν ελκύει τους καταναλωτές, τότε πηγαίνουν οι καταναλωτές σε κάποια website, σε κάποιου τότοπους που είναι όμως παράνομοι. Και όλοι είπαμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή της υποκριτικότητας, αλλά επίσης αυτό θα πρέπει να ισχύσει ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουν υπόψη το κοινοτικό δίκαιο και κυρίως τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όταν συνέταξα την έκθεσή μου, ε, ακολούθησα την προσέγγιση του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εστίασε την προσοχή μου στα εξής. Σε συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο, χρησιμοποίηση καταναλωτών, ε, συνεργασία των κυβερνήσεων, ε, ξέβλημα χρήματος ε, και επίσης ε, λήψη υπόψη του των αθλητικών δρομένων και βέβαια θεωρώ ότι, ότι το κράτος δικαίου ε, είναι ότι κατησχεί μια που και εγώ είμαι νομικός και οπότε θα πρέπει να δούμε ότι εάν θεσπίζουμε κάποιους κανόνες για την ενιαία αγορά τότε κάποια κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να, θα πρέπει να, να, να μην τηρούν αυτού του κανόνε και να υπάρχει ατιμορρησία, γιατί τότε δεν έχει νόημα όμω. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τι διαδικασίε επί παραδιάση. Νομίζω θα πρέπει να γίνουν οι διαδικασίε ταχύτερε και θα πρέπει επομένω να έχουμε ε, σαφέ μήνυμα που να στείλει το Κοινοβούλιο ε, στο ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη ε, να μπορούν να ρυθμίσουν την, την αγορά των τυχαίων παιχνιδιών και θα πρέπει όμως αυτό να γίνεται σύμφωνα στους κανόνες της ιστορικής αγοράς. Επίσης είναι πρωτοφανές, προφανές ότι, θα, ότι όλοι θέλουν να, μοιράζονται τις καλύτερες εμπειρίες, τις καλύτερες πρακτικές και εμείς επομένως είμαστε υπέρ και θα υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν όλη την ίδια ισχύ αλλά θα πρέπει να υπάρξει διάλογος να πάμε σε καλύτερο διάλογο και περισσότερη συνεργασία είτε διμερή είτε πολυμερή ε, για ε, παντού. Οπότε εμείς ως ε, προστασ... επιτρέπωση καταναλωτών θέλουμε να υπάρχει μια καλά ρυθμισμένη ιστορική αγορά ε, που να είναι επίσης ασφαλής για τους καταναλωτές. Εάν δεν έχουμε τέτοια ρύθμιση, τότε έχουμε κάποιους ε, καταναλωτές που οι πιο ευάλωτοι από αυτούς στρέφονται εις προσφορές παρανομές και κάτι το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον ουδενός. Εκεί εστιάζω επομένω ε, τα πράγματα στην έκθεσή μου, αλλά βέβαια έχω καλύψει και τι ιδέε των συναδέλφων για σχετικά με το πώ να αναβαθμίσουμε το σύνολο καταναλωτών. Οπότε έχουμε ε, το θέμα του να είναι έντιμοι οι αγώνε, καθαροί, ε, να μην έχουμε ξύπνημα χρήματο και συμπεράσμα, πρέπει να σα πω κατακλείδη πρόεδρε μια που δεν έχουμε χρόνο, ότι θα κάλυψα τους συναδέλφους, τους σκιοδοσηγητές και επίση θα λάβω υπόψη αυτά τα οποία ο κύριο Υπουργό του θα μα ε, αναλύσει. Uh, Εμεί ευχαριστούμε για την εισήγηση σα, λέει ο Οπότε τώρα θα δώσουμε ε, το λόγο στου δύο εμπειρογνώμονε που έχουμε εδώ για να μα πούν τι γίνεται με την νομοθεσία των τυχερών παιχνιδιών. Πέντε λεπτά έκαστο. Ξέρω ότι δεν είναι αρκετό χρόνο, αλλά έχουν τα σχετικά έγγραφα. Κύριο Σακριάρα, ο οποίο είναι σύμβουλο του Υπουργού Ιστορικών στην Φιλανδία σε σχέση με θέματα διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Και έχουμε επίσης και τον κύριο Φαβιάν Πικάντο, τον ε, Υπουργό του Γιβραλτάρ. Ως πρωτολόγος τον κύριο Υπουργό για πέντε λεπτά. Α, μας έχετε δώσει ένα έγραφο με την ομιλία σας. Thank you very much indeed. Um, I had been told to try and keep it to 10, so all that we'll try and do is speed through... And... Μου είπανε να, να μιλήσω 10 λεπτά, τόσο μπορεί να είναι επιταχύνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δώσατε την ευκαιρία τώρα να έρθω να σας μιλήσω και να σας πω πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα, τι έχουμε κάνει όσον αφορά τα τεπιγραμμικά τυχερά παιχνίδια, τι ισχύει στο Γεβαλτάρ και πώς βλέπουμε το μέλλον αυτού του κλάδου. Όπω γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, έχουμε 30.000 πληθυσμό και μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 40 χρόνια. Και πριν από 40 χρόνια είχαμε αυτό, τέτοια παιχνίδια που ξεκίνησαν και ε, είχαμε τυχερά παιχνίδια που γινόταν το ποντάρισμα με το τηλέφωνο ή με φάξ. Και από την αρχή πριν από 15 χρόνια. Ξεκινήσαμε επομένως ε, την, το αποπόσταση ποντάρισμα που είπαμε ότι θα πρέπει να γίνεται με, με, με, με καθαρού, καθαρούς όρους Και γιατί είπαμε ότι θέλουμε να υπάρχει ε, ποιοτική ρύθμιση. Οπότε γι' αυτό το λόγο τώρα ε, και έχουμε τις κορυφαίες εταιρείε που ήρθαν να εγκατασταθούν εκεί. Από Ηνωμένο Βασίλειο και από παντού. Κύριε Πρόεδρε, αυτός ο κλάδος ε, ανηθεί πάντως σε όλο τον κόσμο και θα συνεχιστεί. Εμείς πάντως, εμείς δίνουμε έγκριση μόνο σε ασφαλείς εταιρείε. Εκείνες που εκτιμούν το, το ότι θα πρέπει το όνομά τους να είναι καθαρό. Αυτό θέλουμε και εμείς. δεν θέλουμε να προλογιστούν αυτέ οι εταιρείε για το κοντάσμα από απόσταση. Ε, θέλουμε να υπάρχει ένα στεγανό σύστημα. Έχουμε επομένω δώσει κάποιες εγκρίσει, κάποιες αδειοδοτήσει. Οπότε αυτές οι εταιρείε τώρα λειτουργούν και εκμεταλλεύονται τα πλέον εκτήματα της ουστικής αγοράς. Βεβαίως όμως εμείς έχουμε θέσει κάποιους περιορισμούς στη λειτουργία που δεν έχει θέσει κανείς. Ας πούμε, εάν ένα κράτος μέλος θεσπίσει κάποια νομοθεσία που ικανοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι ε, αυτό το νομοθέτημα σύντονο προς την συνθήκη, τότε οι, εταιρείε ε, και σε εμά έτσι θα πρέπει να λειτουργούν. Η Ιταλία, Γαλλία, Δανία, Ισπανία έχουν τη δική τους νομοθεσία ούτως ώστε να μην ε, έχουν ε, μονοπόλια και προστατευτισμό, αλλά να υπάρχει ανταγωνιστική. Ε, και οπότε και εμείς τότε είπαμε ότι αυτοί που λειτουργούν σε εμά θα πρέπει να πάρουν και μια άδεια από, τον, το κράτο όπου λειτουργούν και είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλου και όχι μόνο τι εταιρείε που πάνε στην Είμαστε το, το μόνο κράτο που ζητούμε, ζητήσαμε μάλλον από τι εταιρείε ε, να εγκαταλείψουν τη ΣΥΠΑ όταν θεσπίστηκε ένα νομοθέτημα το 2006. Αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη η Επιτροπή σας. Οπότε τώρα ε, είχαμε πάρα πολλές μεγάλες ζημιές από, από διάφορες εταιρείε ε, γιατί έφυγαν από τις ΕΠΑ και όσον αφορά το, το, το, το, το πόκερ ε, ήταν μεγάλε ζημίε γιατί φύγανε από εκεί. Θα πρέπει να σα πω επίση ότι αυτό όμω αποτέλεσε ένα μάθημα το οποίο πήραμε. Και ε, ε, έτσι κινείται η αγορά στη χώρα μα και να σα πω τώρα πώ γίνεται η ρύθμιση και να σα πω τι, τι πρόγραμμα δράση έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά έχουν και την σύγχυση του κ. Φόξ. Πρώτα πρώτα είπαμε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται με τι αρχέ τη τουρκική αγορά και θα πρέπει να κατησχεί πάντα το κράτος ε, δικαίου. Θα πρέπει επομένως να είναι σαφές το δίκαιο, ούτω, αν θέλουμε η αγορά να λειτουργεί καλά. Εάν υπάρχουν κάποια κενά, παραθυράκια στο νόμο, τότε οδηγούμεθα ε, σε, ανασφάλεια, τότε ε, δεν έχουμε την σωστή προστασία του καταναλωτή. Άρα, εάν δεν υπάρχει σωστή δράση για να καλύψει αυτές τις αρχές, τότε συνεχίσουμε να έχουμε το, το, το, το ρίσκο του να ε, στριμώχνονται αυτοί οι οποίοι συμμορφώνονται με το δίκαιο και να ε, έχουν πλεονέκτημα αυτοί οι οποίοι ε, παραβιάζουν τον νόμο. Άρα χρειάζεται συνεργασία μεταξύ επιμυστικών αρχών και κρατών μελών. Οπότε γι' αυτό και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί σε όποιον ενδιαφέρεται για αυτές τις αρχές. Πάντω δεν τα έχουμε πάει καλά μέχρι σήμερα για τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών που πολλέ φορέ δρούν αυτόνομα και δεν συνεργάζονται με τους συνεργούς της άλλα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό δεν είναι υπέρ των, ε, των, των, των καταναλωτών, αλλά έτσι γίνονται τα πράγματα. Οπότε θα πρέπει να λάβετε υπόψη το, το ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και στι ε, χρηματαγορέ. Κοιτάξτε, το Γεβαλτάρ εξορισμού ε, φιλοξενεί ε, τις πιο μεγάλες εταιρείες ε, τυχερών παιχνιδιών ε, με ποντάσμα από απόσταση, αλλά συνεχώς διαπιστώνουμε ότι οι δημιουργικές αρχές δρούν αυτόνομα και γι' αυτό και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα των προσπαθειών σας θα είναι ότι θα ενθαρρυνθεί μεγαλύτερη συνεργασία, περισσότερη συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και επίσης έχουμε δεσμευτεί όσον αφορά πάρα πολύ καλές επιδόσεις μας όσον αφορά τη, τη ρύθμιση των ε, προστατευτικών μέτρων, κάτι το οποίο για όλη την, την Ευρώπη. Έχουμε εμπειρογνωμοσύνη σχετικά και μπορούμε και θέλουμε να μοιραστούμε την εμπειρογνωμοσύνη μας με όλους όσους ασχολούνται με την αγορά με αυτόν τον κλάδο και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, Πρόεδρε, ότι όλες οι εταιρείε του Γιβραλτάρ ε, βοηθούν τις εθελοντικές φιλανθρωπικές οργανώσεις σε σχέση με την υποστήριξη όσων έχουν πρόβλημα με τα τυχερά παιχνίδια και τον εθισμό. Οπότε είχαμε την τρίτη οδηγία κατά του ξεβλήματος ε, ε, χρημάτων, κάτι το οποίο έγινε το 2008. Επίσης, διερευνούμε, εξετάζουμε κάθε καταγγελία ε, καταναλωτή. Έτσι θεωρούμε ότι είναι σωστή η προστασία του καταναλωτή. Επίσης, θέλουμε να ε, υλοποιηθούν οι συστάσεις της Επιτροπής σας. Και επίσης να δούμε τι θα γίνει με τον εθισμό σαν τυχερά παιχνίδια. Είμαι θα εις θέση να, να προωθήσουμε μια κοινή βάση δεδομένων όσον αφορά τους πελάτες των περιοχών αυτών επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το, την τέταρτη προτεραιότητα του σχέδιου δράσης σε σχέση με την απάτη για το ξελινά χρήματος. Εν κατακλείδη κύριε Πρόεδρε, συνεχίζει να ισχύει η δέσμευσή μας όσον αφορά το ότι θα πρέπει να δίνουμε έγκριση μόνο στις πιο σοβαρές εταιρείες εταιρείε που θέλουν να έχουν τεχνολογία, προσωπικό στη χώρα μας και έτσι να μπορούμε εμείς να εποπτεύουμε αυτές τις εταιρείε. Και ε, να μην, χρημα... να μην υπάρχει εταιρική μορφή με τον άνθρωπο ο οποίος ε, ε, δρά κάπου μακριά από την αγορά. Και επομένως θεωρούμε ότι όλοι όσοι έχουν έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι εγκαταστημένοι εκτός από οπουδήποτε άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε φιλοξενήσει επομένω για 15 χρόνια τέτοιε εταιρείε στη χώρα μα και έτσι θεωρούμε ότι υπάρχει ένας τη τη πρακτική, προσθέτει καταναλωτή, ε, κατόξιμονος χρήματο και έτσι θεωρούμε ότι τα κρατημέλη θα πρέπει να ελέγξουν, θα πρέπει να προσέχουν την ε, παράκαμψη του νόμου όσον αφορά την ποντάζουμε από μακριά. εμεί. κάνουμε ε, αυτό το έχουμε κάνει πράξη, το πρέπει να το κάνουν και άλλοι. Και αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι αναγνωριζόμεθα ως ε, ένα σταυροδρόμι για, τις, ε, για το ποντάρισμα του απόσταση, για τυχερά παιχνίδια. Είμαστε η Silicon Valley αυτού του κλάδου και γι' αυτό και έχουμε ελκύσει τέτοιες εταιρείες και καινοτόμες εκεί στο, στο νότιο άκρο της Ευρώπης και θα πρέπει επομένως να είμαστε δημιουργικοί, να μην είμαστε αρνητικοί και θα βλέπει επομένω τα πρότυπα της χώρας μας να ισχύσουν και αλλού. Ε, αυτό το, το πρότυπο του Γιβραλτάρ και το πρώτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να θεωρούνται παράδειγμα προς μίμηση ε, σε όλο τον κόσμο όσον αφορά ε, την νομοθεσία σχετική με τα τυχερά παιχνίδια και θεωρούμε ότι έτσι μπορούμε να πετύχουμε την ανάπτυξη του κλάδου και την προστασία του καταναλωτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφής η πρόθεση να μοιραστούμε τις γνώσεις ο ένας του άλλου και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ε, θα θέλαμε τώρα να καλέσουμε και κάποιον άλλον ο οποίος ε, άμεσα ασχολείται με την ρύθμιση του ζητήματος ε, των στοιχημάτων και των τυχερών παιχνιδιών. Έρχεται από την άλλη άκρη της Ευρώπης, από τη Φιλανδία, είναι ο κύριος Σακάρη Άιρας, ο οποίος είναι σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα τυχερών παιχνιδιών πρέπει να πω στους συναδέλφους ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ξανά το θέμα. Εδώ είναι μόνο το ξεκίνημα της συζήτησης, θα έχουμε και ακρόαση μετά. Ε, δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τον χρόνο μας, αλλά ε, ε, θέλουμε να βοηθηθούμε λίγο, να κατανοήσουμε καλύτερα τις πρώτες ιδέες του κυρίου Φόξ. Κύριε Αίρας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Καλή σας μέρα τα ε, τυχερά παιχνίδια online στην Φιλανδία καλύπτονται από τον νόμο για τα τυχερά παιχνίδια ε, πρέπει να πούμε ότι καλύπτονται όλες οι επιγραμμικές, όλα τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια ε, και επίσης να διαπιστώσουμε ότι τα τυχερά παιχνίδια δεν είναι μια φυσιολογική οικονομική δραστηριότητα. Ε, το σύστημα βασίζεται σε, στο μονοπόλιο τρίν, τριών ε, εταιριών που είναι οι νόμιμοι ας πούμε operators ε, στην Φιλανδία. Μέσω της πράξεως για τα τυχερά παιχνίδια αυτού του νόμου θέλουμε να διασφαλίσουμε τα νόμιμα δικαιώματα όσων συμμετέχουν σε δημόσια τυχερά παιχνίδια. Ε, ή ε, δίνονται πόροι έτσι ώστε να προωθηθεί η υγεία και η κοινωνική ευζοία, ο αθλητισμός, ε, η φυσική δραστηριότητα, η τέχνη, οι δραστηριότητες των νέων, καθώς επίσης και η υπασία και τα παιχνίδια τα σχετίζονται με την, τα σπορ μάλλον που σχετίζονται με την υπασία. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να ελέγξουμε την ανάγκη των παικτών. Ε, και να αποτρέψουμε τον παίκτη από το να αρχίσει να παίζει και να στοιχηματίζει. Ε, η διαδικασία εγγραφής ε, γίνεται πάντα μέσω χρήσης των προσωπικών ηλεκτρονικών τραπεζικών δεδομένων. Θα πρέπει να πιστοποιηθεί ότι είναι ο παίκτης πάνω από 18 χρονών, ότι έχει τραπεζικό λογαριασμό στη Φιλανδία, έχει φιλανδικό άμκα και έχει μόνιμη διεύθυνση στη Φιλανδία πριν ε, ε, ξεκινήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η ταυτοποίηση ε, του πελάτη. Δεν επιτρέπεται κανένα δωρεάν παιχνίδι, ούτε και το λεγόμενο play money game πριν από την επίσημη καταγραφή. Η καταγραφή θα γίνει οπωσδήποτε χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία της, της τράπεζας, του τροπεζικού λογαριασμού, τα οποία τα, τα ε, επίσης ε, ε, πρέπει να πούμε ότι διασφαλίζεται ότι ο κάθε ένας πελάτης θα έχει μονάχα ένα λογαριασμό παιχνιδιού που θα συνδέεται με ένα τραπεζικό λογαριασμό. Ε, θα ήθελα εδώ να σημειώσω και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά ε, τα παιχνίδια online ε, της 15ης 11 του 2011. Στο σημείο 27 αναφέρεται ότι καλεί και ζητά αποτελεσματικές μεθόδους έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της, των τυχερών παιχνιδιών μεταξύ άλλων με τον καθορισμό υποχρεωτικών ορίων που θα βάζει ο ίδιος ο πελάτης. Όσον αφορά την ταυτοποίηση του πελάτη, αυτή γίνεται ε, πάντα επικαιροποιημένα και σε πραγματικό χρόνο μέσα από τα στοιχεία του Εθνικού, Μητρώου, ε, του Εθνικού Δημοσίου Μητρώου. Ε, γίνεται η πιστοποίηση λοιπόν της ηλικία ε, της ε, διεύθυνσης βάση των πληροφοριών, της βάσης δεδομένων των στοιχείων του πληθυσμού οποιαδήποτε αλλαγή είτε στην διεύθυνση είτε στο καθεστώς επιμέλειας και τα λοιπά αμέσως αμέσως ε, ε, αναφέρονται ε, μέσα από την χρήση κιόλας των πιστοποιητικών και των αρχών του e-banking οι πληροφορίες που δίνονται από τον παίκτη ελέγχονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ε, πληθυσμού. Ε, δηλαδή πρέπει να δοθούν ε, ο ΆΜΚΑ, το τελευταίο το, όνομα και το επώνυμο, η μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, η μόνιμη διεύθυνση στο εξωτερικό εάν υπάρχει, τόπους κατοικίας, ηλικίας και επίσης μητρική γλώσσα. Ε, όλοι οι λογαριασμοί των παιχτών ελέγχονται μέσα από αυτό το σύστημα καταγραφής ε, του πληθυσμού και μάλιστα ε, σε τακτική βάση έτσι ώστε είτε παίχτες που έχουν πλέον πεθάνει είτε παίχτες οι οποίοι έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό να αφαιρεθούν από τον κατάλογο των πελατών. Σύμφωνα με την ε, ε, μελέτη του, την τελευταία έρευνα ε, για τον πληθυσμό της Φιλανδίας ο οποίος παίζει βλέπουμε ότι όλο και λιγότεροι είναι αυτοί που ασχολούνται και εν πάση περιπτώσει έχει υπάρξει μείωση του προβλήματος. Ευχαριστώ. Ίσως η κυρία Βιωτικά μπορεί να δει ότι είναι πολύ σχετικά και θα κάνει σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Α ακούσουμε λοιπόν του σκιώδει ηγητέ. Τι λοιπές παρεμβάσεις εάν υπάρξει χρόνος. Ο κύριος Ταραμπέλα, βλέπω ότι ενδιαφέρεται, αλλά πρώτα η κυρία Πιετικά είναι βεβαίως για να ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ και βεβαίως έχοντα υπόψη μου την πίεση χρόνου θα είμαι όσο δυνατόν πιο σύντομη. Καταρχάς ευχαριστώ τον εισηγητή που ξεκινάει τη συζήτηση για την πρόταση παραμένω πεπισμένη ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή συμβαστική λύση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Ένα θέμα με ιδιαίτερη αξία και σημασία. Που θα πρέπει πιστεύω να λύσουμε ανέξατος των πολιτικών επιλογών. Ε, πάντως κάποια θέματα θα ήθελα να τα θίξω εδώ γιατί θα ήθελα να αντικατοπτρίζονται καλύτερα στην έκθεση. Και καταρχάς, γιατί αυτό σχετίζεται πολύ με τη φύση ή τον τρόπο με τον οποίο σταχθεί η έκθεση, ε, θα ήθελα περισσότερες ε, αναφορές στην αρχή ως προς την ε, ιδιάζουσα φύση της χαρτοπεξίας. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι, δεν είναι μια κοινή εμπορική δραστηριότητα. Επομένως, θα ήθελα να υπογραμμιστεί ότι είναι διαφορετικές οι διατάξεις από τις λοιπές διατάξεις εσωτερικής αγοράς, επειδή ακριβώς δεν είναι μια κοινή δραστηριότητα ε, η χαρτοπεξία. Έχει άζους αφήσει όπως και το εμπόριο σιγαρέτων κτλ. Έτσι λοιπόν. Έχουμε μέλημα προστασίας του ατόμου, του ιδιώτη, πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο και θα κάνω τις σχετικές τροπολογίες. Δεύτερον, δεδομένου ότι όπως ακούστηκε εδώ, έχουμε παραδόσεις διαφορετικές στην Ευρώπη, παραδόσεις που θα πρέπει να γίνουν σεβαστές, η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει να καταγράφεται πιο ξεκάθαρα στην έκθεση έτσι ώστε να έχουμε περισσότερη συνέπεια ως προς ε, την χαρτοπεξία τη διαδικτυακή, ενδεχομένως και ανεξάρτητη ε, νομοθεσία, αλλά πάντως με σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας που πρέπει να επιβληθεί και στις ε, σχετικές εταιρείε της διαδικτυακής χαρτοπεξίας. Θα πρέπει να σέβονται και τις εθνικές διατάξεις. ο εντοπισμός ενός λογαριασμού, ο ένας λογαριασμός στον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές και όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πρέπει να καταγράφονται, αλλά ίσως πιο σαφή γλώσσα θα ήταν καλό να έχουμε για να ενισχυθεί αυτό το κομμάτι. Εν όλο, στην έκθεση κρότης μας νομίζω έχουμε ήδη αρκετά καλά στοιχεία. Και από εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε σε βάση. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε θέση σας περιμένω να έχουμε πολύ καλή συνεργασία κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ κυρία Σάλα Ευχαριστώ πολύ και τους δύο μιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Είναι πάντα χρήσιμο να γνωρίζουμε πώς ένα κράτος μέλος έχει ρυθμίσει κάποια κατάσταση. Και το πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι έχουμε πολύ, διαφορε... πολύ μεγάλες διαφορές προς την αντιμετώπιση της διαδικτυακής χαρτοπεξίας ανάλογα με το κράτος μέλος. Πρέπει λοιπόν να το σεβαστούμε αυτό, πρέπει να το σεβαστούμε και για το μέλλον. Και κυρία Πιέτη Κάινεν, νομίζω ε, το σημειώνει ότι χρειάζεται να είναι πιο σαφής αυτή η εικόνα στην έκθεση. Και εγώ θα καταθέσω τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να είναι πιο ε, σαφής η αναφορά στην αρχή της επικουρικότητας και την ανάγκη του σεβασμού προς το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να νομοθετεί και να ρυθμίσει τα ζητήματα αυτά στην επικράτειά του. Όλο το ζήτημα επίσης του πώς ε, μπορεί να τηρείται αυτή η αρχή της επικουρικότητας Και εδώ θα συμφωνήσω με την κυρία Πιετικάρη. Νομίζω ότι χρειάζεται μια διαφορετική διατύπωση. Ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι είναι μια συνήθις οικονομική δραστηριότητα από το διαδίκτυο ή η διαδικτυακή χαρτοπεξία. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι ξεχωριστό. Επίσης, η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών καλά περιγράφεται, θα μπορούσε να βελτιώθηκε λίγο η περιγραφή, αλλά πάντως είναι απαραίτητο να πιεστούν τα κράτη-μέλη για στενή συνεργασία στον τομέα αυτών. Μια σταδιακή διαδικασία ασφαλώς πρέπει να πιεστουν τα κρατη μελη για στενη συνεργασια στον τομεα αυτων μια σταδιακη διαδικασια ασφαλω πρεπει να περιγραφει με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Η δε προστασία των καταναλωτών πιστεύω θα πρέπει να συζητηθεί για το πώς μπορεί να προχωρήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζετε ότι έχουμε πολύ μεγάλο μέλημα για την προστασία του καταναλωτή, κάθε καταναλωτή και κυρίως προστασία από την διαφήμιση υπό κατά τρόπο βέβαια καλύτερο από ό,τι τώρα. Είμαι βέβαια ότι μπορούμε να βρούμε καλές λύσεις και με χαρά περιμένω τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε ότι αναφέρθηκε το όνομα του κ. Κρότσμαν, τον ο Έχει η Επιτροπή μας ιστορία μακρά ως προς την προαγωγή θεμάτων τέτοιων. Περιμένουμε από εσά κύριε Κρότσμαν λοιπόν να μα δώσετε την πείρα σα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλκον. Ευχαριστώ τον κύριο Φόξ για την έκθεσή του. Θα προσπαθήσουμε να τον στηρίξουμε και να ε, τον βοηθήσουμε να ενισχύσει την έκθεση που είναι κάπως περιορισμένη αρχικά. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με διατάξεις που αφορούν την παρέμβαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περίπτωση που η νομοθεσία ενός κράτους μέλους δεν είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, τόσο όσον αφορά το ε, μονοπόλιο, το κρατικό μονοπόλιο, όσο και την απελευθέρωση των αγορών που ε, δεν μπορεί να είναι ε, μονομερείς. Τα, μονοπόλια βεβαίως θέλουν να διαφυλάσσουν τα δικαιώματά τους, αλλά από την άλλη ε, δεν είναι πάντοτε σύμφωνες με τις ε, ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή σχετικές ε, άδειε, Έτσι λοιπόν οι δυνατότητες για διαφήμιση και δραστηριοποίηση των μονοπωλίων εδώ είναι το θέμα της σαφούς διατύπωσης του κειμένου που βλέπω διαφορές μεταξύ του αγγλικού και του γερμανικού κειμένου. Η ασφάλεια του δικαίου επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά την αδειοδότηση, γιατί δεν είμαι βεβαίω ότι, βεβαίως ότι είναι η αδειοδότηση μέσω μιας σύμβασης με τις κρατικές αρχές η λύση. Ε, για τη διοικητική συνεργασία χαιρετίζουμε την ε, πρόθεση για ένα σύστημα ταυτοποίησης των παιχνιδιών, των ε, διαδικτυακών, ε, της διαδικτυακής χορτοπηξίας. Ακούσαμε τώρα τι κάνει η Φινλανδία ως προς την ταυτοποίηση του διαδικτυακού ε, της χαρτοπεξίας της ε, διαδικτυακής ε, είναι κάτι το υποδειγματικό αυτό που κάνει η Φινλανδία. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί ζητάτε επικουρικότητα σε κάτι στο οποίο έχουμε τόσο καλά πρότυπα. Γιατί να μην θέλουμε να κάνουν και τα άλλα κράτη-μέλη το ίδιο καλά ε, την νομοθεσία τους, το, ίδιο καλά όπως η, Φινλανδία. Πρέπει να ακολουθήσουμε το σύστημα της βέλτιστης πρακτικής και όχι να μιλάμε για επικουρικότητα εφόσον στόχος μας είναι δεδηλωμένα προστασία του ε, καταναλωτή, του πολίτη, του νέου από τον κίνδυνο της χαρτοπεξίας. Άρα πρέπει να περάσουμε από τα συστήματα της αδειοδότησης για να αποφύγουμε ή να καταπολεμήσουμε τη μαύρη αγορά, την κρίζα αγορά, ε, την ε, μη ορθή ε, δραστηριότητα τη χαρτοπεκτική στο διαδίκτυο. Ένα σύστημα λοιπόν ενημέρωσης επίσης θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Η ε, περίτη γραφειοκρατία βεβαίως θα πρέπει να αποφευχθεί όσον αφορά τη διαδικασία της ε, ε, αδειοδότησης, ε, εάν ε, παραδείγματι μια δραστηριότητα έχει λάβει άδεια σε ένα κράτος μέλος, τουλάχιστον προς τα τεχνικά τη στοιχεία δεν θα χρειάζεται να περνάει από, θα πρέπει να χρειάζεται να περνάει από την ίδια διοικητική διαδικασία. Κάτι που δεν βλέπουμε επίσης στο κείμενο είναι η καταπολέμηση των παράνομων, δηλαδή των μη αδειοδοτηθισών δραστηριοτήτων χαρτοπεξίας, σε αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Στη δική μου την ε, έκθεση παραδείγματι είχε γίνει αναφορά ως προς την κυκλοφορία χρήματος μεταξύ των μη, αδειοδο... αδειοδοτησών και των ε, αδειοδοτηθησών ε, δραστηριοτήτων, όπου πρέπει να δώσουμε έμφαση προκειμένου να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. φυσικά δεν θα πρέπει οι διατάξει σχετικέ με την αδειοδότηση να είναι τόσο βαριέ και δυσκίνητε ώστε τελικά να σπρώχνουν και τον καταναλωτή στον, ε, στην μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα. Ε, μέλημά μας επίσης ασφαλώς πρέπει να είναι η προστασία του λιγότερο ε, ικανού, του νέου δηλαδή. Ε, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας με μέτρα αναγνώρισης ταυτοποίησης, την υποχρέωση για την ε, αναγνώριση της ε, ή την ε, συμμετοχή μόνο σε ηλικία από μια συγκεκριμένη ηλικία και μετά, απαγόρευση πρόσβαση στο διαδικτυακό χαρτοπέγνιο ή στοίχημα του παίκτη που έχει αναγνωριστεί ως παθολογικός ε, δηλαδή πρέπει να είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνει κακό τελικά στον ε, καταναλωτή που θα συμμετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες. Και βεβαίως, Μάλκομ, δεν χρειάζεται να το πω, ε, δεν πρέπει να μετατρέπεται αυτή η διαδικτυακή χαρτοπηξία σε έναν τρόπο ξεπλήματος παράνομων εσόδων. Έχουμε δει και τα σχετικά με τον αθλητισμό. Είχαμε και μια έκθεση την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερω. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρο. Έχουμε εδώ πέρα ένα εξαιρετό πάνελ με, με του εμπειρογνώμου. Κύριε Πιετικάνη που είχε κάνει έκθεση στο παρελθόν και που είχε βοηθήσει τον κύριο Φόξ και τώρα θέλει. Ε, κυρία Στάιλερ, μπορείτε να. Α, μιλήσετε μετά για να μιλήσει κύριε Ρίλε. Ευχαριστώ και θέλω να ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους δύο μιλητές μας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο παρουσιάσεις που έγιναν. Ο κύριος Φόξ όντως νομίζω ότι είχε πολύ περιορισμένο χώρο για να ε, αναπτύξει όλες τις θέσεις του μέσα σε μια έκθεση. Θα συμφωνήσω με την κυρία Σάλτε Μόντε και την κυρία Πιέτη Κέινεν. Ε, είναι προβληματικό το ζήτημα αυτό. Δηλαδή η τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών που είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντική για μένα αλλά πρέπει να, να εξυπηρετεί κάποιο σκοπό και ο σκοπός αυτός θα πρέπει για μένα να είναι η καταπολέμηση της παθολογικής χαρτοπεξίας και η η παρεμπόδιση της λειτουργίας μιας γκρίζας ή μαύρης αγοράς, παράνομης δηλαδή χαρτοπεξίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό και οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές, οι διατάξεις θα πρέπει να εξεταστούν ε, όχι με, αποκομμένες από το υπόλοιπο πλαίσιο. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Κρότσμαν, σε όλα, εκτός από το ζήτημα της διαφήμισης, γιατί νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιάζον επιχειρησιακό πρότυπο και πρέπει να ε, πούμε ότι και η διαφήμιση έχει εδώ ιδιαίτερη ε, θέση και χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε βεβαίω να αφήνουμε τα κράτη-μέλη να, να υποκρύπτονται πίσω από την ε, επικουρικότητα, γιατί έχουμε εμεί το δικό μα γερμανικό μοντέλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να παρεμποδίσουμε χάρη τη επικουρικότητα τα βήματα για την καταπολέμηση του παράνομου παιγνίου. Γι' αυτό λοιπόν περιμένω και από την ε, δική σας ε, πρόταση να δω τι συγκεκριμένα έχετε προτείνει και αναλόγως να καταθέσω τις προτάσεις τροπολογίας για τον κύριο Φόξ. Γιατί είναι πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα στο Κοινοβούλιο και πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Η Σκιώδης, παρακαλώ, κύριος Γιώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι όσο μπορώ συνόματο. Σε όσα θα σα πω και πρώτα απ' συμφωνώ με κύριε για τι αρχέ οι θα πρέπει να διέπουν αυτήν την ε, έκθεση. Συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Επίση θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι συνέπειε, ε, ας πούμε στην παραγραφωτερία Τη εκθέσεις που λέει ότι τα μονοπόλια των παιχνιδιών δεν θα πρέπει να μειώνουν τις ευκαιρίες και θα πρέπει εμένα υπό προποθέσει να ε, σύρονται οι εταιρείε αυτών των δικαστηρίων. Ε, ναι, να μην μειώνονται οι, οι ευκαιρίε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη χορμή του νόμου με αυτά τα μονοπόλια. Τουλάχιστον αυτό ισχύει για τη χώρα μου. Ένα, αυτό. Δεύτερον, αυτού του είδου το, το, η γραφειοκρατία που λέμε, αυτό το διοικητικό βάρο ούτω το δεν θα πρέπει να είναι αυτός σκοπός. Οπότε, εν προκειμένου, θα πρέπει πάντοτε να, να αιτιολογείται η, η κάθε ρύθμιση. Τώρα, ε, εδώ πέρα, θα πρέπει να δούμε αν έχει αρκετή η Επιτροπή, θα πρέπει επομένω να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά, όσον αφορά την ρύθμιση ε, του, του, του, των τυχερών παιχνιδιών μέσω ίντερνετ. Άρα, για πέστε μας τι τεκμηρίως έχετε, από πού προέρχεται. Έχω λάβει εδώ κάποια στοιχεία, αλλά θα ήταν χρήσιμο να μας λέγατε περισσότερα, διότι στην έκθεση έχετε πει ότι η απαγόρευση θα οδηγήσει σε περισσότερο παράνομο στοιχηματισμό. Δεν και δεν έχω πιστεί τώρα. Υπάρχουν κάποια που έχουν παραλείψει το ρόλο των τραπεζών όσον αφορά τις πληρωμές, με τα ε, συναλλαγές, με τα παράνομα site, ε, η διαφήμιση, η σχετική νομοθεσία, πώς θα εφαρμοστεί παντού για τις εποπτικές αρχές είναι δυνατόν να τις ε, να υπάρχουν σε όλα τα κατημέρια και υποχρεωτικά να συνεργαστούν και τέλος το βασικό θέμα που είναι το ξύλμα χρήματος, το ξέρουμε αυτό ε, είδατε πώς, πώς κατέληξε τώρα να απειλείται η Ευρωζώνη γιατί το ξύλμα χρήματος ε, συνδέεται πάρα πολύ και με τον παράνομο και με τον νόμιμο στοιχηματισμό και τυχερά παιχνίδια. Μα είπαν τη γνώμη του όλοι και ο και από ό,τι μπορείτε να δείτε. Ωστόσο τώρα έχουμε σιγά σιγά εδώ την προσέλευση ε, όλων που θα λάβουν μέρο στην επόμενη ακρόαση. Άρια, ε, Ραβάλ, ε, Ταραμπέλα κλπ. Θέλετε τώρα να μιλήσετε μισό λεπτάκι ή να τα πείτε όλα μαζί με την ευκαιρία της ακρόασης που θα ακολουθήσει. Τώρα, τώρα μισό λεπτό. With Mr. Tarabella, and this clock will start now. Bon, ben, je serai bref, Président, et je vous quitterai juste après, non pas pour échapper au feu des questions, mais je... τώρα θα σα τα πω. Όχι, όχι, όχι, δεν, θα πρέπει να, να φύγω να πω κάπου άλλο. Τέλο πάντων, με, με, με έχει σοκάρει η έκθεση Fox, διότι. Όχι, όχι, με, με όλου συμφωνούμε προ το Γιβραλτάρ. Δεν κάνουμε έκθεση για το Γιβραλτάρ, αλλά έχουμε και το Μονακό και το Λιχτενστάιν, τα οποία ανοίγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε κύριε εκπρόσωπε του Γιβραλτάρου θα πρέπει όντως να εκμεταλλευόμαστε την, ε, την ιστορική αγορά αλλά όμως εσείς δεν την ωφέλει τόσο πολύ και βλέπω ο κύριος Ντεγιόν του αρέσουν οι μελέτες επιπτώσεων Θα γίνει μελέτη επίπτωση όσον αφορά την απασχόληση που εσείς δημιουργείτε στη χώρα σα και καταστρέφετε σε άλλε. Και επίσης να δούμε τι γίνεται με τα έσοδα. Γιατί υπάρχουν κάποιε εταιρείε ε, που αφορούν ε, κάποια λαχεία. όμω. την άλλη μεριά η υποστήριξη οικονομική το, του αθλητισμού, το, των, ε, των, των πρακτορείων, των παιχνιδιών και διάφορα νομικά πρόσωπα και δίκτυα αυτών που υπάρχουν. Ε, ο, τι κάνετε εσεί τώρα δεν δίνει τίποτα στους άλλους και, και εσείς όλοι ε, ελκύετε όλες τις καλύτερες εταιρείε και λέτε ότι όμως βοηθάτε κάποιες, κάποιες φιλανθρωπικές εταιρείε. Καλά πρέπει να φύγω κύριε Φόξ. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Ναι, ναι, ήμουν πάρα πολύ καλός μέσα σας. Κύριε Φιέλνερ, για εσάς όμως θα είμαι πιο αυστηρό. Μάλκομ, σε ευχαριστώ. Ναι, ναι, θα είμαι σύντομο. Ευχαριστώ και τον Άσλι Φόξ, είναι πάρα πολύ καλή αυτή η έκθεση και είναι, αποτελεί μια σωστή συνέχεια τη της έκθεσης ε, και επίση να δούμε ότι όντω θα πρέπει να έχουμε νομοθεσία για τέτοια παιχνίδια αλλά όχι σβάρο του καταναλωτή και τη προστασία του καταναλωτή. Αυτό είναι το, το, το δίδαγμα μας γιατί θα, θα, θα έχουμε το δικαίωμα, την υποχρέωση να ελέγχουμε τον διασυνοριακό χαρακτήρα, ιδίω στου αγορά των καταναλωτών. Επομένω, η ερώτησή μου ακριβώ αφορά τον το, το, το Φιλανδό κύριο. Εάν κανεί είναι εθισμένο στα τυχερά παιχνίδια και εάν κανεί κάποια στιγμή έχει ένα φωτεινό διάλειμμα, πώ μπορεί να αυτοεξαιρεθεί, μπορεί να αποχωρηθεί, να, κάποιο να κόψει κάθε είδου ποντάρε με τυχερό παιχνίδι στη Φιλανδία ή να το απαγορεύουν το να παίζει, να παίζει, να παίξει σε κάποια χώρα, αλλά μπορεί να πάει άμα του να παίξει αλλού σε άλλη ας πούμε, έχει κόψει τη Φιλανδία και να πάει να παίξει στην, στην Αγγλία. Ε, αυτό είναι θέμα προστασία των κανοτών, κάτι το οποίο είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αναφερθώ μονάχα στην προστασία των καταναλωτών, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, αλλά παρόλα αυτά να, ε, παρουσια... να αναφέρω μάλλον τρία άρθρα το άρθρο 10 όπου διαπιστώνεται όπου για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να υπάρξει μια ε, σωστή προσφορά τυχερών παιχνιδιών. Εγώ δεν θέλω πλήρη απαγόρευση, αλλά πιστεύω ότι η προστασία των νέων ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να αναφερθεί ε, ή τουλάχιστον να αναφερθεί με μεγαλύτερη ρόμη. Άρθρο 12. Όντως χρειαζόμαστε μελέτες αντικτύπου, επιπλέον μελέτες, ας πούμε το Ινστιτούτο Ανάλυσης των Εξαρτήσεων έχει κάνει έρευνα όσον αφορά τα καζίνο στα κράτη-μέλη και νομίζω ότι οι συστάσεις που έχουν απορρεύσει από την έρευνα αυτή καλό θα ήταν να αναφερθούν. Τέλος, άρθρο 15. Το ανέφεραν ήδη κάποιοι συνάδελφοι όσον αφορά την διαφήμιση δηλαδή. Στην έκθεση γίνεται αναφορά ε, μονάχα στην απατηλή διαφήμιση, αλλά κοιτάξτε, εμείς νομίζω ότι εδώ πρέπει να μιλήσουμε για διαφήμιση που θα είναι κοινωνικός ορθή. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, λέει ο πρόεδρος, θα έχουμε και άλλη δυνατότητα και ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα θέματα αυτά. Τέλος, ο κύριος Αρίας. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Ακούσαμε πολλά πολλά πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν για να τονιστούν περισσότερο στο έγγραφο στην έκθεση Fox. Εγώ θέλω να σταθώ σε ορισμένα από αυτά τα σημεία όπως η επίλυση των προβλημάτων για την προστασία του καταναλωτή, του χρήση, η προστασία των δεδομένων επίσης, όπως το ανέφερε Μάλκο, ε, σύμφωνα με το φιλανδικό πρότυπο, νομίζω είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα μια που το φιλανδικό μοντέλο είναι αξιόλογο και θα πρέπει επομένω να λάβουμε υπόψη τα δεδομένα και την δημοσίευσή τους. Επίσης άλλο ζήτημα είναι η προστασία των ανηλίκων. Uh, now, um, Mr. Fox, can you, um, Κύριε Φόξ, μπορείτε πολύ σύντομα ε, να ολοκληρώσετε Ευχαριστώ βέβαια και τον ε, κύριο Τέμικ που είναι εδώ από την ε, ε, Κομισιόν. Είμαστε λίγο καθυστερημένοι, λίγο αργοπορημένοι, δεν πειράζει. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Έγραψα εδώ πολλές σημειώσεις. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους. Πάντως, να ευχαριστήσω τους δύο καλεσμένους μας που ήρθαν εδώ έτσι ώστε να μας εκθέσουν την πραγματογνωμοσύνη τους. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους. Δεν θα απαντήσω γιατί δεν θέλω να απαντήσω σε μερικούς και να αφήσω κάποιους άλλους που έθεσαν ερωτήματα ε, να αφήσω τα ερωτήματά τους αναπάντητα. Θα μιλήσουμε ξανά για το θέμα αυτό σε ένα-δυο μήνες. Πάντως σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά στο διάλογο. Τροπολογίες 4 Απριλίου. Κάποιοι συνάδελφοι και εσείς το είπατε ότι ε, η, ε, πρόκειται εδώ για ίδιας πρωτοβουλίας έκθεση και πρέπει να είναι σύντομη θα υπάρξουν ε, πολλές τροπολογίες, ε, είμαι βέβαιος. Ξέρω ότι συνεργάζεσαι στενά και με τους ε, εισηγητές, τους σκιώδες εισηγητές. Πάρα πολύ ωραία. 24-25 Απριλίου θα λάβει χώρα η επόμενη μεγάλη συζήτηση. Θα προβλέψω με αρκετό χρόνο έτσι ώστε να έχουν όλη τη δυνατότητα να εκφραστούν με την ησυχία τους ε, για το θέμα αυτό και ίσως ε, να έχουμε και την Κομισιόν στην επόμενη συνεδρίασή μας ε, να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ και τους καλεσμένους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Και να σας πω ότι και ο λόγος του, και η παρέμβαση του κυρίου Ρικάρντο θα είναι στον ιστό τοπό μας. Πάρα πολύ ωραία. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερησία διατάξεως που προβλέπει ακρόαση. Κοιτάξτε παρακαλώ, πολύ ησύχως δεν καταλήψετε την αίθουσα εάν δεν προτίθεστε να παραμείνετε ε, για να παρακολουθήσετε την ακρόαση έτσι ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς θόρυβο. Θα ξεκινήσω λοιπόν τώρα τη συζήτηση όσον αφορά την έκθεση για την οποία εισηγητής θα είναι ο κύριος Μάντερ, τον οποίο και καλωσορίζω. Το θέμα λοιπόν είναι η απλοποίηση της μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος εντός της νέας αγοράς έχουμε την ε, πρόταση. Θα ακούσουμε όμως ε, πρώτα μια παρουσίαση της Επιτροπής ε, η οποία θα παρουσιάσει την πρόταση. Ο κύριος Μάτσεκ θα εκπροσωπήσει εδώ την Επιτροπή. Υπάρχει και ένα θέμα με, τον, με τη μελέτη αντικτύπου Θέλουμε να δούμε επίσης το κατά πόσον ε, μπορεί κανείς ε, να ε, διευκολύνει την ταξινόμηση μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος στα πλαίσια μιας καλά οργανωμένης ενιαίας αγοράς. Θα ζητήσω από τον εισηγητή συντόμως να εισαγάγει την συζήτηση και μετά θα δούμε και τους εμπειρογνώμονες, θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες που έχουμε καλέσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μάντερς. Ναι, πρόκειται για ένα από τα 20 ε, πιο σημαντικά προβλήματα για τα οποία προσφεύγουν και ε, οι καταναλωτές και για τα οποία έχουμε παράπονα από τους καταναλωτές. Εδώ η πρόταση είναι καλή και ελπίζουμε ότι μαζί με τους σκιώδεις ε, θα καταφέρουμε να βρούμε έναν κανονισμό που θα ικανοποιεί ε, τους ε, πολίτες. Έχουν προσκληθεί διάφοροι εμπειρογνώμονες ε, για να μας δώσουν παραδείγματα ε, για την ενδεχόμενη βελτίωση του κανονισμού ε, για τρόπους με τους οποίους όλη αυτή η κατάσταση να γίνει πιο εύκολη για τις κυβερνήσεις αλλά να διευκολύνει ταυτόχρονα και τους πολίτες. Εάν όλα πάνε καλά ε, πιστεύουμε ότι η βιομηχανία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων θα βρει μια νέα άνθηση γιατί βρίσκεται σε μαρασμό τώρα ε, και νομίζω ότι γενικώ η αγορά ε, του αυτοκινήτου θα πάρει τα πάνω της, κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα αυτή η αγορά. Απ' την άλλη πλευρά Νομίζω ότι βελτιώνοντας την οικονομία στο σύνολό της ε, θα ικανοποιήσουμε και το, τους πολίτες μας. Θα ζητήσω λιγότερο χρόνο έμπειρο εμπειρογνώμονα έτσι ώστε να έχουμε πιο ζωντανή συζήτηση ε, ξέρετε ποια είναι η άποψή μου, να έχουμε καλές πληροφορίες, ε, να τις χρησιμοποιήσουμε καλά έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την οδηγία. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ε, στάση σας. Ναι, έχουμε απομονώσει, έχουμε ταυτοποιήσει μάλλον τα 20 πιο σημαντικά σημεία προβληματισμού για τους πολίτες και αυτό το θέμα των αυτοκινήτων είναι ένα από τα προβλήματα. Θα καλέσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, να μας ε, πει δύο λόγια όσον αφορά ε, το background της πρότασης και μετά 10 λεπτά για τον κάθε εμπειρογνώμονα θα δούμε. Θα δούμε και θα παρακολουθούμε και την ώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ που προσκαλείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας παρουσιάσει την έκθεση που ήδη έχει υιοθετηθεί. Εδώ και ένα χρόνο περίπου. Πέρσι τον Απρίλιο. Προσπαθούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίσει ο πολίτης όταν θέλει να μεταφέρει την ταξινόμηση του οχήματός του σε μια άλλη χώρα. Πρόκειται για τον τομέα ο οποίος παρουσιάζει και τις περισσότερες καταγεγραμμένες ε, προσφυγές ε, ως προς το ε, ως προς το πρόβλημα της μη εναρμόνισης της αγοράς. Προσπαθούμε λοιπόν να διευκολύνουμε και να κάνουμε πιο απλή τη ζωή των πολιτών, οι οποίοι πολύ συχνά αντιμετωπίζουν πολυάριθμες διαδικασίες, διαδικασίες που διαφέρουν σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη και έτσι η πρότασή μας πιστεύουμε ότι έχει σημασία μεγάλη για την καθημερινή ζωή του πολίτη αλλά και του επιχειρηματία για τη λειτουργία της επιχείρησης. Διότι πολλοί είναι οι εμπλεκόμενοι πιστεύω στην υπόθεση αυτή φορείς αυτοί δηλαδή οποίοι θα είχαν ενδιαφέρον να συζητηθούν τα θέματα αυτά. Γιατί λοιπόν υπάρχει το πρόβλημα αυτό, γιατί έχουμε την διασυνοριακή αυτή, τα συνοριακά αυτά προβλήματα και πολύ σύντομα και πολύ συχνά γιατί διαμαρτύρονται οι πολίτες γιατί όλες αυτές οι παραβιάσεις της νομοθεσίας και γιατί χρειάζεται να εξετάσουμε τόσο συχνά τις ε, διαδικασίες και διατάξεις που ισχύουν. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι πολύ συχνά το ότι δεν είναι σαφές το πού θα πρέπει να γίνει η ταξινόμηση του οχήματος. και ότι τα κράτη-μέλη συχνά δεν αναγνωρίζουν ταξινόμηση, δεν αποδέχονται δηλαδή την είσοδο ενός ε, οχήματος που έχει ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος. Δηλαδή συχνά ε, σταματούν το όχημα και ο ε, ιδιοκτήτης του αντιμετωπίζει προβλήματα, ερωτήσεις ε, σε σχέση με την χώρα ταξινόμησης, συνθήκες ταξινόμησης κτλ. Άρα αυτό θα το, θα το αντιμετωπίσει η πρότασή μας. Εν συντομία για το ιστορικό της πρότασης, είχε προτείνει η Επιτροπή να εναρμονιστεί ο φόρος ή το τέλος καλύτερα ταξινόμησης διότι αυτό ουσιαστικά είναι και η βάση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης. Το, ε, το κύριο αίτιο. Δυστυχώς όμως αυτή η πρόταση ε, αντιμετώπισε προσκόμματα και δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Προσπαθούμε λοιπόν να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα σε σχέση με, την, με το τέλος ταξινόμησης. Νομίζω ότι δεν έχει κανείς αντίρρηση ως προς το τέλος ταξινόμησης ε, σε ένα κράτος άλλο από το κράτος προελεύσεως, απλώς ε, πρόβλημα αποτελεί η πληθώρα νομοθεσιών, γραφειοκρατικών διαδικασιών κτλ. που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να ε, γίνει ταξινόμηση σε ένα άλλο κράτος. Προσπαθούμε να εναρμονίσουμε τις ε, διατάξεις και να τις απλοποιήσουμε και να περιορίσουμε το γραφειοκρατικό βάρος, φόρτο. Πώς θα το κάνουμε αυτό, προσδιορίζοντας το πού θα πρέπει να γίνει η ταξινόμηση ή αντίστροφα υπό ποιου όρου μπορούν να ζητήσουν, να απαιτήσουν την ταξινόμηση οι αρχέ του κράτου μέλου. Δηλαδή, κοιτάμε την ρύθμιση από τη σκοπιά περισσότερο του πολίτη και όχι τη αρχή. Και λέμε ποιο είναι το κράτο το οποίο μπορεί να ζητήσει την ταξινόμηση ενό οχήματο. Αντί να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη την υποχρέωση σε κάποιε συγκεκριμένε συνθήκε, εφόσον συντρέχουν κάποιε συγκεκριμένε συνθήκε, να ταξινομούν. Διατυπώσει. Προσπαθούμε να μειώσουμε τι διατυπώσει για τη διαδικασία τη ταξινόμηση και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών ενημέρωσης μεταξύ των κρατών μελών. Στο στόχο λοιπόν, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε το στόχο αυτό, έχουμε ε, εξετάσει διαφορετικές εναλλακτικέ. Ε, παραδείγματι την, αρχή, την απλή αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών που προκύπτει από την ε, συνθήκη. Ε, με την ε, επιπλέον τήρηση των διαδικασιών περί παραπομπής ή παραβάση. Ωστόσο με πολύ μαζικές ε, μετακινήσεις πολιτών, είτε για επαγγελματικούς είτε για οικογενειακούς λόγους, ίσως είναι δύσκολο να τηρηθεί αυτή η αρχή. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να γίνεται μία μόνη ταξινόμηση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη μία ταξινόμηση στο πρώτο κράτος μέλος ή με μια ενιαία ταξινόμηση για τα οχήματα που θα ίσχυε για ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος. Αλλά και πάλι αυτή η επιλογή για λόγους που έχουμε αναπτύξει πιο διεξοδικά στο κείμενό μας δεν έγινε δεκτή. Ε, και έτσι φτάνουμε σε μια πρόταση συμβιβαστική η οποία προσπαθεί να εξισορροπήσει τα διάφορα συμφέροντα τα διάφορα και ποικίλα συμφέροντα, με θετικό αντίκτυπο για την ζωή του πολίτη. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να μετακινηθεί ένα όχημα ε, από τη μία χώρα στην άλλη. Θα είναι πολύ, πολύ πιο ευχερής η αγορά ή η πώληση ενός οχήματος από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Θα είναι πολύ πιο εύκολο ο καθημερινός βίος των ε, μεθοριακών των εργαζομένων στις παραμεθόριες περιοχές και θα είναι πολύ πιο ευχερής η μετακίνηση ε, μεταξύ μιας κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας όταν ε, ο ενδιαφερόμενος έχει ένα όχημα και θέλει να μπορεί να ε, μετακινείται από τη μία στην άλλη κατοικία χωρίς προβλήματα. Για τις επιχειρήσεις θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για τους αντιπροσώπους πώληση μεταχειρισμένων για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, οχημάτων και για τους πελάτες τους. Επίσης οι εθνικές αρχές θα δουν απλούστευση του ε, έργου τους, του φορτού εργασίας, όπως επίσης θα περιοριστεί η εγκληματικότητα σχετική με τα ε, οχήματα, ε, γιατί θα υπάρχει μία μόνο ταξινόμηση αναγνωρισμένη μεταξύ κρατών μελών, θα είναι πιο ευχερή η επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Κύρια στοιχεία της πρότασης. Όπως είπα, η οδηγία, η πρόταση κανονισμού στηρίζεται στην αρχή ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν ταξινόμηση εφόσον ο κάτοχος του πιστοποιητικού ταξινόμησης έχει τη συνήθη κατοικία του στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους. Δηλαδή, βασική αρχή ότι ε, έχουμε το τεκμήριο ότι καθής χρησιμοποιεί το όχημα του στο κράτος το οποίο έχει τη συνήθη κατοικία του. Δεν κοιτάμε τη χρήση τόσο, αφήνουμε κατά μέρο την αρχή τη χρήση, την προσέγγιση με βάση τη χρήση, γιατί αυτό είναι πολύ περίπλοκο, και κοιτάμε απλώ να χρησιμοποιήσουμε ένα σαφέ ε, κριτήριο, όπω τη συνήθη κατοικία του πολίτη. Άλλωστε αυτό το καταγράφει πολύ πιο λεπτομερό στο άρθρο 3 της προτάσεως, όπου ορίζουμε το τι νοείται ως συνήθις κατοικία. Είτε έδρα επιχείρησης, είτε κατοικία φυσικού προσώπου. θεσπίστε μια απλουστευμένη ε, διαδικασία επαναταξινόμησης και έτσι, εάν ο κάτοχος του πιστοποιητικού ταξινόμησης μετακινηθεί, μετακομίσει για λόγους προσωπικούς, οικογενειακούς, επαγγελματικούς, Μπορεί να διατηρήσει το όχημα λοιπόν, να μετα κομίσει σε άλλο κράτος μέλος, περίπτωση κατά την οποία θα χρειαστεί να γίνει επαναταξινόμηση μέσα στο εξάμεινο που ακολουθεί την άφηξή του στο νέο κράτος μέλος. Θα χρειαστεί στην περίπτωση αυτή να ε, προσκομίσει αποδεικτικά ότι είχε ταξινομηθεί σε άλλο κρατός μέλος το όχημα, να προσκομίσει το πιστοποιητικό ταξινόμησης. Οπότε οι αρχές ταξινόμησης του νέου κράτους μέλους θα μπορούν χάρη στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών να συλλέξουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. δεν θα χρειάζεται επιπλέον να κάνει κάτι επιπλέον για την επαναταξινόμηση στο κράτος προελεύσεως ο ή από το κράτος προελεύσεως καλύτερα ο πολίτης, γιατί αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά με την αυτόματη ε, ε, επικοινωνία των αρχών. Επομένως δεν θα επιβαρύνεται περισσότερο ο πολίτης. Στην περίπτωση αγοράς οχήματος, διάφοροι κανόνες, διαφορετικοί κανόνες, ε, δίνεται ε, ένα περιθώριο 30 ημερών, εφόσον είναι κανείς ήδη εγκατεστημένος και έχει συνηθικατική σε ένα κράτος μέλος ε, και εισάγει από άλλο κράτος μέλος ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα. Αυτό το κάνουμε και με μια ε, ειδική διάταξη για ταξινόμηση που θα σας αναφέρω σε λίγο. Απλουστευμένες διαδικασίες επαναταξινόμησης που συνεπάγονται επιπλέον και άλλες διατάξεις απλουστευμένες, δηλαδή λέμε ξεκάθαρα πού θα γίνεται ο τεχνικός έλεγχος ή η επιθεώρηση του ε, οχήματος. Δηλαδή η συνήθιση διαδικασία θα είναι η επιθεώρηση, η αυτοψία στο όχημα να μην χρειάζεται, γιατί θεωρούμε και πιστεύουμε ότι θα το δεχθούν και οι ειδικοί, ότι είναι πολύ πιο σημαντική αναγνώριση αμοιβαία παρά η αυτοψία. Βέβαια, κατά περίπτωση θα περιτρέπονται και οι αυτοψίε, όταν έχει σοβαρή ζημιά, υποστεί το αυτοκίνητο, το όχημα ή αν υπάρχει σοβαρό λόγο ε, να θεωρηθεί ότι οι τεχνικές διατάξεις ε, βάσει των οποίων έχει καταχωρηθεί σε άλλο κράτος μέλος ε, το όχημα δεν είναι ευθεγραμμισμένε με αυτέ του, του νέου κράτου, του κράτου υποδοχή. Άρα οι αρχέ του κράτους λίγο πολύ θα πρέπει να αποδέχονται την αμοιβαιότητα ή την αναγνώριση των τεχνικών διαδικασιών που ισχύουν ε, και της επιθεώρησης που ισχύει στο άλλο κράτος μέλος, αν και μπορεί να υπάρξει και άρνηση από την αρχή ε, του κράτους υποδοχής για την επαναταξινόμηση. Η πολύ σημαντική διάταξη που ανέφερα νωρίτερα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών ταξινόμησης. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα, απλουστεύει την διαδικασία επαναταξινόμησης Αναφέρθηκα επίσης σε προσωρινή ταξινόμηση ή πιστοποιητικό. Η προσωρινή ταξινόμηση θα πρέπει να καλύπτει το χρονικό εκείνο κενό μεταξύ της αγοράς σε ένα κράτος μέλος και της μεταφοράς σε ένα άλλο κράτος μέλος του οχήματος, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου ε, οχήματα μεταχειρισμένα πολλούνται σε νέο ιδιοκτήτη, χάνουν το πιστοποιητικό που είχαν στο πρώτο κράτος μέλος και τότε προκύπτει το ερώτημα πώς μπορούν να μεταφερθούν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σύστημα προσωρινή ταξινόμησης που επιτρέπει εντό 30 ημερών την ολοκλήρωση των ε, διατυπώσεων στο νέο κράτος μέλος και μία πρόταση η οποία ε, προσπαθεί να διευκολύνει τη χρήση από τον επαγγελματία του οχήματος, εταιρείε που έχουν ε, διανομή, συντήρηση ή ε, υπηρεσίες δοκιμής οχημάτων με ιδιαίτερα κριτήρια που είναι και οι επαγγελματικές δεξιότητες, ικανότητες και η καλή έξω μαρτυρία θα μπορούν να προχωρούν σε αυτή την χρήση ε, υπό τις ειδικέ συνθήκες που ισχύουν για την ειδική αυτή επαγγελματική ε, ταξινόμηση. Τι άλλο. Αυτό είναι το περιεχόμενο της προτάσεως. Ελπίζουμε να υιοθετηθεί στα τέλη του 2013, το πολύ αρχάς του 2014 και ο κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μέσα σε ένα έτος από τη στιγμή της έγκρισης του. Προβλέπονται επίσης διατάξεις για κατεξουσιοδότηση πράξης και τα στερόχρονα από τη θέση ισχύ θα γίνει μια αξιολόγηση ώστε η Επιτροπή να εξετάσει πώ λειτουργεί αυτό ο κανονισμός και αν φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, είναι αποτελεσματικό όπως θα θέλαμε. Σας ευχαριστώ θερμά και είμαι στη θέση σας για οποιασδήποτε ερωτήσει. Uh, ευχαριστώ πολύ που μας περιγράψατε και μας ε, δώσατε λεπτομέρειε για την πρόταση της Επιτροπής αν μου επιτρέψετε, τις ερωτήσεις θα τις ε, κάνουν οι συνάδελφοι αργότερα. Θα δώσουμε τον χρόνο πρώτα απ' άλλου στους ε, άλλους ε, ομιλητές, οι οποίοι δεν θα έχουν πάνω από 10 λεπτά, αν έχετε τη δυνατότητα. Έχουμε όλοι ένα αντίγραφο των βιογραφικών σας και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με πολύ σύντομες παρουσιάσεις. Ε, θα δούμε πρώτα απ' όλα ε, την ε, άποψη των εκπροσώπων των οδηγών και της αυτοκινητοβιομηχανίας κατά κάποιο τρόπο. Καλωσορίζω την Κλόντια Μέη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημόσια ευρωπαϊκή πολιτική της ΑΝΤΑΚ. Δέκα λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ως ενεγνωρισμένη Ένωση Καταναλωτών με 18 εκατομμύρια μέλη, η, Ευρω... η Γερμανική Οδική Βοήθεια, ADAC παρακολουθεί τα προβλήματα και τις ε, προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τα αντιμετωπίσει. Χαιρετίζουμε λοιπόν ρητά της Προσπάθειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την πρόταση για την ε, νέα νομοθετική πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να τοποθετηθούμε. το νομικό τμήμα της ΑΝΤΑΚ ε, λαμβάνει καθημερινά περί τις χίλιες προτάσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, προσφυγές για νομικά θέματα σχετικά με την κινητικότητα, εκ των οποίων 20% έχουν να κάνουν με το διεθνές δίκαιο της κυκλοφορίας της οδικής κίνησης δηλαδή και έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια ε, γενική επισκόπηση και ιδέα για το τι συμβαίνει και ιδιαίτερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Γερμανία. Πολλά είναι τα ερωτήματα των μελών μας σχετικά με τις υπερσυνοριακές αδειοδοτήσεις και ταξινομήσεις. Προβλήματα προκύπτουν κυρίως όσον αφορά την αγορά ενός αυτοκινήτου σε κράτος μέλος, άλλο από αυτό της ε, κατοικίας ή αλλιώς ε, σε περίπτωση μετακόμιση από το ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο. Χρειάζεται λοιπόν μια απλουστευμένη μορφή για ταξινόμηση πέραν των συνόρων και για κάποιον ο οποίος θέλει να ε, ζει σε ένα κράτος μέλος και να μετακομίσει σε ένα άλλο, σε κάποιον που ζει κοντά στα σύνορα αλλά εργάζεται από την άλλη μεριά των σύνορων, σε έναν πολίτη που ενδεχομένω έχει μια εξοχική κατοικία σε ένα άλλο κράτος μέλος και ιδιαίτερα την Ισπανία όσον αφορά τους Γερμανούς, έχουμε τέτοια ζητήματα. Και ξεκινώ λοιπόν με το πρόβλημα της αγοράς αυτοκινήτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΑΝΤΑΚ υποστηρίζει τα μέλη της και όσον αφορά ακόμα και τα γλωσσικά προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν κατά την αγορά ενός αυτοκινήτου εκτός από την ε, Γερμανία. Όταν ένας αγοραστής λοιπόν θέλει να αγοράσει ένα όχημα στο εξωτερικό, ε, τίθεται συχνά το ερώτημα του πώς μπορεί να μεταφέρει το όχημα αυτό στην ε, Γερμανία με πολλές δυσκολίες, πολύ συχνά, διότι βασικά θα πρέπει να έχει το έγγραφο ή το πιστοποιητικό εξαγωγής το όχημα αυτό και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο αγοραστής είναι ότι δεν είναι αναγνωρισμένο το σχετικό πιστοποιητικό εκτός Γερμανίας, εφόσον, το έχει, εφόσον βρίσκεται στην Γερμανία και δεν μπορεί να ε, αποκτήσει τέτοιου είδους πιστοποιητικό εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει και σχετικό πιστοποιητικό κατοικίας. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε προβλήματα τα οποία σημαίνουν και πολύ μεγάλο κόστος αλλά και περιπλοκές νομικές. Πολύ συχνά ε, βρίσκουν μια λύση οι αγοραστές με τη μεταφορά αυτού του πιστοποιητικού, αλλά ουσιαστικά είναι παράνομη και σε σχέση με το γερμανικό δίκαιο, αλλά και σε σχέση με το δίκαιο άλλων κρατών. Τη σχετική μέθοδο την έχει απαγορεύσει πρόσφατα η Ιταλία με αποτέλεσμα πολλές φορές να φτάσουμε και σε δημεύσεις αυτοκινήτων αλλά σημαντικά πρόστιμα μέχρι ε, και 800 ευρώ πρόσφατα το Φεβρουάριο πρόστιμο που προέκυψε λόγω της οδήγησης χωρίς την ε, απαιτούμενη αδειοδότηση ή την ε, οδήγηση χωρίς ασφάλιση. Αυτό μόνο και μόνο επειδή οι Ιταλικές αρχές δεν αναγνώριζαν το σχετικό γερμανικό έγγραφο. Βεβαίω ε, η ΑΝΤΑΚ προσπαθεί πάντοτε να δώσει συμβουλές τους ε, στα μέλη της, να ε, βοηθήσει στην ταχεία κάλυψη του προστίμου κτλ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει το σχετικό ε, πιστοποιητικό, ένα πιστοποιητικό μεταφορά του οχήματο από το ένα κράτο στο άλλο, ώστε ε, να υπάρχει και η αναγνώριση από τι ασφαλιστικέ εταιρείε και με μία μόνο ε, προσέγγιση που θα αφορά μόνο μία αρχή. Η διαδικασία τώρα. Η διαδικασία για την αδειοδότηση στο εξωτερικό έχει πολλέ, για την ταξινόμηση δηλαδή ενό οχήματο στο εξωτερικό, έχει πολλά προβλήματα πολύ συχνά, ιδιαίτερα για αυτού οι οποίοι ζουν στο ένα κράτο αλλά εργάζονται σε κάποιο άλλο κράτος και ιδιαίτερα για όσους Γερμανούς έχουν σε άλλο κράτος μέλος ε, κατοικία δευτερεύουσα για τις διακοπές τους αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και γλώσσας και γραφειοκρατικά. Η διαδικασία λοιπόν για τους αλλοδαπούς είναι πολύ δύσκολη από ό,τι παρατηρούμε. Ε, συχνά αναγκάζεται ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει σε μία ε, σε ένα γραφείο εξυπηρέτησης ιδιωτικό που πρακτορεύει αυτές τις διαδικασίες και σε εκ τούτου κοστίζει πολύ περισσότερα χρήματα. Που όμως ε, μπορεί να συνεπάγεται και αν δεν τηρηθούν σωστά οι διαδικασίες και πολύ σημαντικά πρόστιμα για τον κάτοχο. Γι' αυτό καλούμε να εισαχθούν διαδικασίες ταχείες, απρόσκοπτες, μη ε, και να μην υπάρχει διαφορά μεταξύ του ενός κράτους και του άλλου, του, του κράτους ταξινόμησης και του κράτους ε, εγκατάστασης. Ε, ο προσδιορισμός του κράτους κατα... ταξινόμησης λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος, διότι η αρχή της αρχής ταξινόμησης έχει πολύ μεγάλη σημασία δεν είναι σαφές εάν θα προσδιορίζεται η ε, χώρα της ε, συνήθους διαμονής ή κατοικίας ή η χώρα της χρήσεως ενός οχήματος. Μεταξύ Γερμανία και Αυστρία, Αυστρίας, παραδείγματι, παρατηρείται το πρόβλημα ότι αν κάποιο Γερμανό συχνά δουλεύει και ταξιδεύει με το αυτοκίνητό του στην Αυστρία, θα είναι μάλλον υποχρεωμένο, ακόμα και η μόνιμη κατοικία του είναι στη Γερμανία, να ταξινομήσει στο αυστριακό σύστημα το όχημά του. Η συνήθιση λοιπόν κατοικία είναι μια σωστή προσέγγιση. Αν και μπορεί σε ορισμένε μεμονωμένε περιπτώσει να οδηγήσει σε σημαντικέ δυσκολίε. Και λόγω τη υψηλή κινητικότητα που έχουμε στην Ευρώπη, θα πρέπει τόσο οι επαγγελματικές, η επαγγελματική προσωπική δεσμοί σε διαφορετικά κράτη-μέλη ενός προσώπου να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδορισμό ενός ορισμού ο οποίος δεν θα δημιουργεί δυσκολίες στην ε, ταξινόμηση. Επίσης, όταν θέλει να ε, θέσει τέλος στην ταξινόμηση ένα ε, πολίτη για ένα αυτοκίνητο το οποίο όμω πλέον δεν βρίσκεται στο κράτο τη αρχική ταξινόμηση, θα έχει πρόβλημα ε, την, την ανάγκη να επανέλθει, να επαναφέρει το αυτοκίνητό του στην, αρχική, στη χώρα τη αρχική ταξινόμηση για να ολοκληρώσει εκεί τις διαδικασίες. Εδώ δεν υπάρχει λοιπόν ε, ρύθμιση και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια απλή διαδικασία περάτωσης της ταξινόμησης, κλεισίματος ταξινόμησης. Επίσης πολύ σημαντικό και εν συντομία στα άρθρα 5 και 6 της προτάσεως του κανονισμού έχουμε τις προϋποθέσεις δυναμή των οποίων τα κράτη-μέλη μπορεί να αρνηθούν ή να απορρίψουν την ταξινόμηση ή επαναταξινόμηση. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν δεν προκύπτει απόδειξη για ε, υποχρεωτική ασφάλιση, ότι υφίσταται υποχρεωτική ασφάλιση, η ελέγχιστη ασφάλιση του αυτοκινήτου. Και τελευταίο σημείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αιτιολόγησή της ε, δηλώνει ότι είναι ελεύθερα τα κράτη-μέλη να ορίσουν τις διατάξεις σε σχέση με, την, ε, με τον ε, κανονισμό και την ταξινόμηση και ότι θα πρέπει να κάνουν προσπάθειες για την προσαρμογή σε μια κοινοτική ρύθμιση. Ζητήματα και φορολογικού χαρακτήρα και άλλα πιστεύουμε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί συχνά ο πολίτης είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση επαναταξινόμησης να καταβάλει νέο τέλος ταξινόμησης από το ένα κράτος μέλος στο άλλο δεν υπολογίστε δηλαδή στην ε, προσμέτρηση του δεύτερου τέλους ταξινόμησης ότι έχει ήδη καταβληθεί ένα τέλος σε άλλο κράτος μέλος. Και... Παρά την θετική αξιολόγηση της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα θέλαμε συμπληρωματικά να πούμε ότι χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σήμα και δεύτερον, πρέπει η καταξινόμηση να γίνεται με σαφεί και πρακτικού ορισμού Και τρίτον, η άδεια και η επαναταξινόμηση να γίνεται συνδεδεμένη με τον σεβασμό του δικαιώματο τη υποχρέωση. καλύτερα για ασφάλιση του οχήματο. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε κύριε Μέη γιατί τηρήσατε ακριβώ το όριο των 10 λεπτών. Και τώρα μας μιλήσει ο κύριος Τζον Λούις. Τζον Λούις είναι εκπαιδευτικός διευθυντής τη ε, Ένωση των ε, εταιριών ενοικιάσεως οχημάτων στην Βρετανία και επίσης ε, εκπροσωπεί τον φορέα του, του, της για την Ευρώπη, ιδίως ε, όσον αφορά τέλος πάντων τα, τα ενοικιαζόμενα οχήματα, για να μας πει τη γνώμη του επαγγελματιών του κλάδου, τι γνώμη έχουν όσον αφορά τι επιπτώσει αυτού του νομοθετήματο. Το πολύ 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ εγώ κύριε Πρόεδρε και σα ευχαριστώ πάρα πολύ διότι μα επιτρέψατε να έρθουμε εδώ και να σας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας για αυτό το θέμα αυτό. Συγχαρητήρια για τα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα. Σήμερα σας μιλώ ως ε, επικεφαλής ε, του Lease Europe. Να σας πω πρώτα πρώτα τι είναι ο φορέας μας. Είναι η Ομοσπονδία των ε, Εθνικών Ενώσεων που εκπροσωπούν τη χρηματοδοτική μίσθωση και την ηλικία αυτοκινήτων μιλούμε για 43 χώρες, 2.000 εταιρείες, οδογικές μίσθωσης και για να δείτε τι, ακριβώς ε, ποιες είναι οι διαστάσεις ε, του ρόλου μας στην αγορά σήμερα ε, τα μέλη μας 14 εκατομμύρια ε, αυτοκίνητα και επίσης επενδυλμετικά οχήματα 5,6 εκατομμύρια. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι επιπτώσει για τον κλάδο μας, για τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Θεωρούμε ότι θα υπάρξουν και διάφοροι φραγμοί ε, σαν ε, επιπτώσει του νομοθετήματος κακές για το καταλωτή. ξεκινω Ξεκινώ. Πρώτα-πρώτα, θα ήθελα να δούμε τι γίνεται με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων προς μια κατεύθυνση όπως ονομάζονται. Ε, έχουμε όλο ένα και μεγαλύτερη ζήτηση από πλευρά καταναλωτών σε σχέση με το ότι θέλουν να διώσουν αυτοκίνητο και να πάνε κάπου, διασύρονται κάποια σύνορα και να μην επιστρέψουν. Και αυτό είναι ιδίω πρακτικό για ε, Κάποιε οικογένειε που θέλουν να πάρουν ένα πολυμορφικό αυτοκίνητο ή να βάλουν μέσα όλους τα πράγματα, τα, τα μπαγκάζια κλπ. αντί να πάρουν ε, αυτοκίνητο ή ταξί. Πάντως, οι δυσκολίε μα είναι ότι δεν μπορούμε να ξανανοικιάσουμε το αυτοκίνητο στη χώρα προορισμού. Οπότε έχουμε ε, παραδείγματα κατά τα οποία έχουμε δει τι έχει γίνει ας πούμε στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας και οπότε το θέμα είναι ότι πρέπει να επαναπατριστεί το αυτοκίνητο. Αυτό ε, βέβαια συνεπάγεται κάποιο κόστος, οπότε και η συναλλαγή αυτή γίνεται πάρα πολύ ασύμφορη. Οπότε ο αναπατρισμός κοστίζει και αυτό πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική λύση. Αν επομένω ε, θεσμοθετηθεί ε, αυτή η πρόταση που είπαμε θα επιτρέψει να είναι δυνατόν να ξαναμισθώσουμε το όχημα στην χώρα προορισμού, χωρίς να χρειάζεται επαναπατρισμός. Ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται με επιπλέον φραγμούς, είναι ότι δεν μπορούμε να ε, νοικιάσουμε αυτοκίνητα επομένως διασυνοριακά. Ε, μιλούμε τώρα για τις διακοπές, σε Ισπανία και σε Νότια Γαλλία. Επομένως θα πρέπει να διπουργήσει και αυτά ώρα για να τα ταξινομεί για να ε, ε, σύνοχνο το διάστημα, αλλά ούτε αυτό συμφέρει γιατί μιλούμε τώρα για την περίοδο του καλοκαιρινή των δύο μηνών. Μας είπαν για εξάμεινο οι συνάδελφοι που το λόγο προηγουμένως. Τότε θα μπορούσαμε τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται αρκετά, δηλαδή αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται από επαγγελματίε αλλά όχι στι διακοπέ, δεν μπορούσαμε αυτά να τα πάμε στην Νότια Ευρώπη. Οπότε θα είχαμε τα αυτοκίνητα που θέλουμε για να καλύψουμε την ε, θερινή περίοδο. Ε, τελικά, όπω και για τα ξενοδοχεία, έχουμε εδώ θέμα ζήτηση και προσφορά. Οπότε έτσι μπορούμε να έχουμε πιο ανταγωνιστικού όρου, ε, μπορούμε να καλύψουμε την ε, ζήτηση. Να δείτε τώρα έχω ένα γράφημα που θα σας ε, δείξω να δείτε πώς πάει η ζήτηση. Οπότε έχουμε επομένως τα, την αναταξινόμηση και το σχετικό κόστος, αλλά επίσης ε, κάθε χρόνο πάρα πολλά αυτοκίνητα 34 ετών και έχουν μέχρι και 100.000 ε, μίλια στο κοντέρ, οπότε αυτά τα οχήματα ε, είναι, προέρχονται από χρηματοδοτικές μισθώσεις και είναι σε αρκετά καλή κατάσταση το πρόβλημα είναι ότι μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση αλλά όμως η μετακίνηση διασυνοριακά δεν συμφέρει γιατί ακριβώς θα πρέπει να γίνει επαναταξινόμηση γιατί είναι ακριβώς αυτή η φραγμή τεχνολογική που μας το πρωί ακριβώς το πρέπει να γίνουν κάποιες επιθεωρήσεις ε, προβλήματα συμβατότητας για τους τεχνικούς ελέγχους. Ε, τα πιστοποιητικά συμβατότητας θα πρέπει να μεταφραστούν ε, στη γλώσσα του κράτους προορισμού, οπότε έχουμε διάφορα παράπονα από την αγορά μεταχειρισμένων θα ήθελαν να μπορούν οι έμποροι μεταχειρισμένων να τα μετακινούν διασυνοριακά, να καλύψουν τον καταναλωτή, κάτι το οποίο σήμερα είναι πάρα πολύ ακριβό και χρονοβόρο. Οπότε, αν γίνεται, να σας κλείσω δύο, δύο λεφτάκια εδώ πώς πάει η, ε, η ζήτηση. Σε αυτό το γράφημα βλέπετε επομένω έχουμε αυτή την γραμμή. Βλέπετε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πιο ακραία από τις άλλες χώρες, αλλά βλέπετε τι γίνεται ανά τρίμηνο. Οπότε ακριβώς για αυτή την περίοδο ε, της υψηλής ζήτησης να δίνεται να έχουμε μόνο για εκείνη διαθέσιμα αυτοκίνητα. Αν έχουμε όμω απλούστερε διαδικασίε ταξινόμηση και αναταξινόμηση, μπορούμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στην εκμίσθωση αυτοκινήτων σε αυτή την περίοδο. Επίση, έχουμε και κάποιε ε, άλλε καταγγελίε και παράπονα, τα οποία αφορούν ε, πρώτα-πρώτα τι εταιρείε χρηματοδοτική μίσθωση που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους σε άλλη χώρα από την αρχική χώρα ταξινόμησης. Οπότε ε, αυτό μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα με αυτό το εξάμεινο το οποίο αναφέρθηκε ως προθεσμία. Βέβαια, η περίοδος της ορματοδικής μίσθωσης έχουν σχέση με τους όρους ταξινόμησης στην αρχική χώρα. Οπότε νομίζω ότι τα τεχνικά ζητήματα μπορούν να επιληθούν εύκολα. Αν και υπάρξει κάποια βασική ρυθμίση νομοθετική. Κάτι άλλο τώρα που αφορά το πώ έχει η νομοθεσία. Ε, θα μπορέσουμε να μεταγίνουμε τα χήματα αν περάσει αυτό το νομοθέτημα και επίση στη χώρα προορισμού μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε γιατί θεωρώ κύριε Πρόεδρε ότι νομίζω καλύψαμε πάρα πολύ καλά που οι προλαλήσαντε τα τεχνικά ζητήματα και τον υπόλοιπο χρόνο που μα μένει μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πιο επικοδομητικά σε απαντήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Πάρα πολύ σαφέ αυτό για όλου εμά που δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τι οικονομικέ λεπτομέρειε. Γιατί είμαστε εδώ πελάτε, αλλά πρέπει να ξέρουμε γιατί γίνεται στο περιθώριο. Έχουμε τώρα τους δύο τελευταίους ομιλητές αυτής της πρώτης, ε, του πρώτου τμήματος και θα ήθελα να μας ε, μιλήσουν για κάποια ευρύτερα ζητήματα τα οποία άπτονται της ε, ασφαλείας των πολιτών. ορίζω λοιπόν τον Πίτερ Βάντερ Έντερ, Program Manager στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ασφάλειας και τον λέων Βαν Ντεν Λάρ ε, ο οποίος είναι Business Development ε, Manager και ProDrive BV ε, στο Brainport στην Ολλανδία. Έχουμε εδώ λοιπόν την ώρα του Brainport με τους δύο μήνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μιλάω πάρα πολύ καλά. Η φωνή μου είναι λίγο βραχνή σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Με καλέσατε κύριε Πρόεδρε για να μιλήσω μαζί με τον Λεόν στη ε, για το ζήτημα της ασφάλειας και, το, το, και της αυτοκινήτων. Εμείς συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα για το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης των ε, πινακίδων των αυτοκινήτων. Ε, εμείς δουλεύουμε στο Brainport Development Εκεί συμμετέχουν και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και με τον τρόπο αυτό ε, το Ολλανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ε, για την Ασφάλεια ε, μπορεί να δουλέψει πολύ καλά. Κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό ε, να ε, έχουμε συνεργασίες ε, με στόχο την καινοτομία, όπως ας πούμε εδώ που μας απασχολεί το ζήτημα της αυτόματης αναγνώρισης των πινακίδων των αυτοκινήτων, όπου οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ αστυνομία, κυβέρνησης, υπουργείων, εισαγγελία, πανεπιστημίων, επιστημονικών φορέων, business partners κτλ. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προτείνουμε στους επενδυτές οικονομική προσέγγιση θέμενη αξία. και οι εταίροι βεβαίω ε, μπορούν ε, να έχουν το, καλύτερο, το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Εμείς αναπτύσσουμε διάφορα προγράμματα ασφάλειας, ας πούμε την βιομηχανική ε, ασφάλεια, την ασφάλεια μάλλον στα βιομηχανικά και τα επιχειρησιακά πάρκα, την ασφάλεια στα το εσωτερικό ε, ε, δακτύλιο των πόλεων, επίσης ε, το secure lane για τα parking κτλ. Θα συνεχίσει ο Λεόν. Καλημέρα, λέγομαι Λέον Βάναντερ Λάρ, είμαι Business Development Manager ε, σε μια εταιρεία που ασχολείται με τα ηλεκτρονικά και με τις ε, ε, κάμερες παρακολούθησης και θα σας πω κάποια στοιχεία όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις για την εξ αναγνώριση. δουλεύουμε και εμείς στο Brainport, έχουμε μια νέα τεχνολογία, αυτή είναι μια μηχανή φωτογραφική η οποία έχει αισθητήρε 20 megapixels δηλαδή 20 φορές μεγαλύτερη λεπτομέρεια ε, στα πλαίσια των ε, καμερών που υπήρχαν μέχρι τώρα στους ε, δρόμους. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να πιάσει κατά κάποιο τρόπο η κάμερα αυτή ή όλα τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στο δρόμο με μεγάλη σαφήνεια εικόνας. και νομίζω ότι με αυτήν την ε, φωτογραφική μηχανή είναι κανείς ε, πάρα πολύ εύκολο να διαβάσει ε, με μεγάλη ανάλυση και σαφήνεια τις πινεκίδες των αυτοκινήτων. Βεβαίως... Το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα φωτογράφησης των οχημάτων όχι μόνο τη μέρα αλλά και τη νύχτα, με λίγο φως δηλαδή. Ε, λοιπόν, ε, ε, εδώ σας δείχνω στα αριστερά την συνήθεια εικόνα των συμβατικών καμερών. Έχουν αυτό το rolling shutter όπως λέγεται, ενώ με την καινούρια κάμερα έχουμε το global shutter με πολύ καθαρότερη εικόνα παράδειγμα για το πώς μπορείτε ας πούμε να πάρετε φωτογραφίες σε διάφορες λωρίδες κυκλοφορίας. Βλέπετε πώς γίνεται Αυτή είναι μια εικόνα, θα έπρεπε κανονικά να είναι κινούμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε σε θέση ε, να κάνουμε ταινίε, αν θέλετε με αυτήν την, ε, ε, με την εικόνα να συμπεριλάβουμε εικόνα και της πινακίδας αλλά και του οδηγού ε, του αυτοκινήτου, ε, ε, εικόνες δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς όπως αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών. Εδώ βλέπετε νυχτερινή μορφή, πώς είναι η κατάσταση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέρα και νύχτα για την επιβολή προστήμων για υπερβολική ταχύτητα βλέπετε τη διαφορά ανάμεσα στην κάμερα την καινούρια αριστερά και δεξιά τη συμβατική κάμερα και άλλες ε, ε, ε, κάμερες οι οποίες είναι σταθερές αν δείτε ας πούμε δεν φαίνεται καλά η πινακίδα με τις ε, συνήθεις συμβατικές σταθερές ε, κάμερες ενώ με την καινούρια μπορεί κανείς ε, να πάρει όλα τα στοιχεία που θέλει με μεγάλη σαφήνεια το, ακόμα και το βράδυ. Ε, και εδώ βλέπετε ότι παρότι τα φώτα είναι αναμένα και η φωτογραφία είναι ακριβώς, πέφτει ακριβώς πάνω στα φώτα ε, και με την κοινή κάμερα δεν είναι σαφής η εικόνα, παρόλα αυτά στην απάνω εικόνα με την καινούργια κάμερα ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αναγνώρισης της πινακίδας. και επομένως με τον τρόπο αυτόν και αυξημένη ασφάλεια υπάρχει και μικρότερος αριθμός καμερών μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ο εισηγητής από την Επιτροπή Μεταφορών δυστυχώς πρέπει να φύγει. Ε, θα τον ξαναέχουμε και αργότερα μαζί μας. Uh, um, ναι, καλύτερα που γύρισε γιατί θα σε χρειαστούμε. Έχουμε και τον Ρόρι Οκόνορ, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, της ομάδας εργασίας της Προεδρίας. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε σήμερα να του δώσουμε το λόγο, αλλά ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι η Προεδρία εργάζεται πάνω στο ε, ζήτημα αυτό. Πριν από ένα χρόνο περίπου αποφασίσαμε ότι ε, ε, έπρεπε και το Συμβούλιο να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό ε, και είδαμε ότι και το Συμβούλιο ξεκίνησε. Βεβαίως καλό θα ήταν να συντονίσουμε λίγο τα προγράμματά μας και τα χρονοδιαγράμματά μας. Λοιπόν, τέσσερι, τέσσερα λεπτά για ερωτήσεις από τους Σκιόδης και άλλους. Είμαι και εγώ σκιώδηση τη. θα θέσω και λοιπόν και εγώ αργότερα μια ερώτηση. Ε, ε, ε λοιπόν, Άντριο Φάμπ από, το, ε, από τους σοσιαλιστές λέει ο πρόεδρος ναι ναι εντάξει εντάξει έκανα κάποια λαθάκια, δεν έχει σημασία. Η κυρία Ρούλε από τους Πράσινους, εγώ από τη δική μου ομάδα. Η κυρία Ρούλε είναι σταθερή στη θέση του σκιώδους, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θα τεθούν ε, οι ερωτήσεις και θα δώσω και τη δυνατότητα στους ομιλητές μας να απαντήσουν αν το επιθυμούν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστώ για, την πολύ, για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Θα θέλω να πω καταρχά ότι το σου ότι είναι παρόν εδώ το ΑΝΤΑΚ, η μεγαλύτερη ένωση καταναλωτών Ευρώπη, έχει να κάνει. Ε, έχει να αποδείξει ότι πολλοί είναι οι πολίτες ε, του οποίου άμεσα αφορά το ζήτημα τη ταξινόμηση των οχημάτων και ευχαριστώ ιδιαίτερο στο ΑΝΤΑΚ που ε, με τόσο επικοδομητικό τρόπο υποστηρίζει τι προτάσεις. Θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αιτιολογήσει, γιατί στο άρθρο 6 της προτάσεως της έχει μια μια μηνιαία προθεσμία, δηλαδή τέσσερι εβδομάδε συγκεκριμένα, για την μεταφορά τη ταξινόμηση. Η κυρία Μάη τη Αντάκ μας λέει ότι αρκούν δύο εβδομάδες και συμφωνώ σε αυτό. Άρα Ρωτώ την Επιτροπή γιατί θεωρεί ότι χρειάζονται οι τέσσερις εβδομάδες στο άρθρο 6. Δεύτερον, Πρόεδρε, υπάρχει περίπτωση από, Ευρωπαϊκή, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής το, η διαδικασία του άρθρου 8 να ε, επιτρέψει και συμμετοχή των των κατασκευαστών αυτοκινήτων ε, στη διαδικασία και στις εργασίες ε, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα. Επίσης έχει στήσει ο κύριος Καράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι εδώ παρόν σήμερα, να είναι η ασφάλιση υποχρεωτική, η παρουσίαση της προσκόπηση δηλαδή πιστοποιητικού ασφαλίσεως, υποχρεωτική για την ε, μεταταξινόμηση ή αναταξινόμηση, πράγμα το οποίο δεν προβλέπεται στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Χάρμπορ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ε, για το θέμα της ασφάλισης. Με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ η Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς έχει προαγάγει, ανέκαθεν προάγει τα συμφέροντα των καταναλωτών και ιδιαίτερα στην προσωρινή μεταφορά ταξινομήσεως που πάντοτε μας, βρίσκει, μας φέρνει αντιμέτωπους με το πρόβλημα της ασφάλισης. Πρέπει λοιπόν αυτό να προβλεφθεί και στον κανονισμό αλλά και στην ε, ε, οδηγία για τα οχήματα με κινητήρια. Κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, προσκεκλημένους μας. Και άκουσα επίσης και τον προηγούμενο αγορητή του ΕΛΚ. Ναι, αυτό που είπε θα το έλεγα και εγώ, γιατί πρόκειται για κάποιο δύνατο σημείο που έχει η πρόταση. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι θέμα τελικά δημοσίας ασφάλειας. κάτι να σας πω σε σχέση με, με, με, τα, με τα κταίω, τη, σχετικά πιστοποιητικά τους, το, το, ότι κανείς ε, μπορεί να πάει όπου θέλει να κάνει τον τεχνικό. Γιατί ε, επ' αυτού δεν ε, ασχολήθηκα με την έκθεση. Και επίσης και για αυτό το εξάμεινο κατά το οποίο μπορούμε να κάνουμε την επαναταξινόμηση. Οπότε Ε, αυτό αποτελεί κάποιο είδου εισόδημα για τα κράτη. Αλλά με τη νέα πρόταση βέβαια το βάρος θα το φέρει η δημόσια διοίκηση. Ας πούμε, το, η διεύθυνση του Υπουργείου Σιωνιών πρέπει να ασχοληθεί, αλλά τώρα θα έχει έξτρα δουλειά. Για, οπότε για πέστε μας. Τι ισχύει στα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάλυψη από τον προπολογισμό. Πολύ ενδιαφέρον. Επίσης και σχέση με το leasing τη χρηματοδοτική μίσθωση. Είναι κάτι το οποίο καίει τους ε, ψηφοφόρους μας. Ας πούμε τότε που είχαμε την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία, ο κόσμος ε, θεώρησε ότι αντί για το αεροπλάνο μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο για να επιστρέψει αφού το νοικιάσει. Θα πρέπει όμως να διευνηθούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και ζητώ συγγνώμη που δεν είναι περισσότεροι εξημών εδώ για να σας ακούσουν. Πάντως το θέμα αυτό το εντοπίζει η Επιτροπή μας πάρα πολύ σοβαρά και επίσης είναι θετικό το ότι έχουμε εδώ και εκπρόσωπο της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ. Κύριε Ρίλη, θέλω το λόγο. Όχι, να σας πω τώρα και εγώ τα εξή. Θα ήθελα να πω κάτι όσον αφορά αυτό που μας είπε ο κύριος Λούις, δηλαδή τη δυνατότητα των χρηματοδοτικών ε, εταιριών, των εταιριών leasing τέλο πάντων, να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητα φέροντας τα από κάποια άλλη χώρα για να τα εκμισθώσουν. Άρα θα πρέπει να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο βασικά είναι ιστορικό κάθε χώρας. Είναι θέμα της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Μας είπατε ότι τα κράτη-μέλη έχουν πάρει κάποιους περιορισμούς και δεν μπορούν να σας αφήσουν, έτσι, δεν σας αφήνουν να χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί σε άλλη χώρα. Άρα, η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής θα σας λύσει τα χέρια. Θα μπορείτε να αναταξινομήσετε το αυτοκίνητο για να το χρησιμοποιήσετε. Να μου φαίνεται βαλωματική αυτή η λύση. Θα πρέπει να γίνει κάτι πιο ριζοσπαστικό να πει κανεί στα κρατημέλη δεν τηρείται την οδηγία για τις υπηρεσίες. Δηλαδή μπορεί να, να σας βοηθάει στη δουλειά σας η εταιρεία, αλλά δεν είναι η καλύτερη λύση. Ένα αυτό που να σας πω. Το άλλο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς θα έχουμε τα θέματα αναγνώρισης τεχνολογίας, αλλά επίσης ε, να έχουμε περισσότερα φωτογραφικά στοιχεία να δούμε το σύστημα πώς θα είναι στεγανό για θα μιλήσουμε αργότερα ε, για το έγκλημα, για την ασφάλεια Κύριε Μάντες έχετε και εσείς ερώτηση Σας ευχαριστώ όσον αφορά την τελευταία σας ερώτηση Κάλεσαν τους καλύτερους ε, εμπειρογνώμονες, γιατί ο κόσμος φοβάται ότι εάν είναι πάρα πολύ απλό να παραταξινομηθεί ένα αυτοκίνητο, θα έχουμε πρόβλημα με τα κλεμμένα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κάποιου επαρκούς ελέγχου. Και γι' αυτό και καλέσαμε τον κόσμο για να εξηγήσουν το πόσο έχουμε συστήματα ελέγχου. Επίσης, είναι και θέμα ελέγχου του ιδιωτικού βίου. δεν θέλουμε από τη μία μεριά επομένω να κυκλοφορούν κλεμμένα αυτοκίνητα, αλλά από την άλλη θέλουμε την προστασία του ιδιωτικού βίου επίση. Σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μα είπε ο κ. Γκόρκα ότι χρειαζόμαστε κάποια ρύθμιση πανευρωπαϊκή. Και θα τα πούμε στο δεύτερο τμήμα της ε, ακρόασης. Θέλουμε μια βάση δεδομένων πανευρωπαϊκή. Οπότε, οι φωτογραφίες που παίρνουν στους δρόμους ε, είναι δεδομένο να τις διαβάσει κανείς άμεσα για να δούμε αν κάποιο αυτοκίνητο είναι κλεμμένο ή να δούμε επίσης κατά πόσον το αυτοκίνητο ε, είναι σύντομο, σύντομο με την νομοθεσία. Κύριε Πάρκινς, γιατί θα επανέλθουμε σε αυτό. Όχι, με τον κύριο Γκόργα θα αρχίσουμε τις απαντήσεις. Και κατόπιν ανάβουμε με τη σειρά το λόγο οι υπόλοιποι κύριοι του πάνελ για να απαντήσουν. Γκόργα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις στους ομιλητές. Θα τις με τη σειρά. Πρώτη ερώτηση για τις τέσσερις εβδομάδες για την ταξινόμηση. Όντως, διαφέρει από κράτος σε, μέλος, σε άλλο κράτος μέλος η κατάσταση. Δεν υπάρχει δηλαδή μία συνήθις περίοδος μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η ταξινόμηση. Σε άλλες είναι δύο, σε άλλες είναι τέσσερις ή περισσότερες εβδομάδες. Εμείς έχουμε ορίσει τις εβδομάδες προκειμένου να αφαιθεί αρκετός χρόνος για όποιον αγοράζει αλλού το όχημα. Και στην περίπτωση προσωρινής ταξινόμησης πάλι για να μπορέσει να καλυφθεί το ε, διάστημα αυτό από την προσωρινή ταξινόμηση στη μόνιμη. Να έχει ο κόσμος στη διάθεση του αρκετό χρόνο και να αισθάνεται ασφαλής ότι προλαβαίνει να ολοκληρώσει τις διατυπώσεις χωρίς ε, πίεση. Για την ασφάλιση. όντως δεν περιλαμβάνεται εδώ ως ε, προϋπόθεση για ταξινόμηση ή ασφάλιση. Μπορεί να αποτελέσει βέβαια λόγο άρνησης από πλευράς του κράτους μέλους της επαναταξινόμησης. Πάντως δεν είναι και συνήθις ε, προϋπόθεση στα κράτη-μέλη η ασφάλιση. Δηλαδή δεν απαιτείται πάντα να προηγηθεί της ταξινομίας ως η ασφάλιση μερικές φορές την ε, ε, έπεται. Και εμείς δεν θέλουμε με την αναρμόνιση αυτή να επιβάλλουμε στις χώρες για τις οποίες δεν απαιτείται η προηγούμενη ασφάλιση να γίνεται αυτή προκαταβολικά πριν από την αναταξινόμηση. Υπάρχουν άλλες διατάξεις, χωριστές διατάξεις που αναφέρατε κι εσείς που έχουν να κάνουν με την οδηγία για την ασφάλιση των οχημάτων με κινητήρα και αυτές πρέπει να τηρηθούν, αλλά δεν θεωρούμε ότι απαιτείται να αναφερθούν δωρητά. Για το εξάμεινο. Και τη δημοσιονομική διάσταση τα έσοδα δηλαδή των κρατών μελών. Όπω είπα, δεν επηρεάζει αυτή η πρόταση την φορολογία, την επιβολή τέλου. Η περίοδο την οποία ε, χορηγούμε εδώ ω περιθώριο για να μετακινηθεί ένα αυτοκίνητο δεν έχει συνέπεια ω προ το πότε θα επιβάλλει το κράτο την καταβολή του τέλους. Αυτή την αρμοδιότητα τη σεβόμαστε. και νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα αρμοδιότητας των κρατών μελών. Το περάρτημα. Το περάρτημα καταγράφει στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η βάση δεδομένων και που πρέπει να είναι και προσβάσιμα στα άλλα κράτη κατά την επαναταξινόμηση ενός οχήματος υποχρεωτικά στις τις περιπτώσεις το κατά πόσον πληρούνται ή μη οι προϋποθέσεις είναι ακόμα, το πώς επαληθεύεται δηλαδή η πληρώση των προϋποθέσεων είναι ακόμη υποσυζήτηση. Είναι κάτι το οποίο θα ακολουθήσει την ε, έγκριση και τα τεχνολογικά, τα τεχνικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μέη. Χωρίς μικρόφωνο. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στην ε, περίοδο αυτή των τεσσάρων εβδομάδων. Θα δείτε ότι και οι τέσσερις εβδομάδες και οι έξι μήνες καταγράφονται στην πιο αναλυτική μας ε, παρατήρηση. Είναι υπερβολικά γενναιόδορη αυτή η περίοδος των τεσσάρων εβδομάδων για μας. Δύο εβδομάδες νομίζουμε ότι αρχούν, αρκούν για μια συγκεκριμένη αναταξινόμηση προκειμένου να αποφευγόνται και οι καταχρήσεις. Το ίδιο και για το εξάμεινο. Η μείωση σε τρεις μήνες της περίοδου αυτής νομίζω πάλι θα έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των καταχρήσεων. Γιατί βάσει δεδομένων αναφερθήκατε νομίζω στην διακοπή της καταχώρησης ή την επιστροφή πυρακίδων Θα ήθελα λίγο να μου εξηγήσετε την ερώτησή σας, την παρατήρηση σας μάλλον, και επίσης για την απόδειξη ασφάλισης, πιστοποιητικό ασφάλισης. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τα κράτη-μέλη τα οποία απαιτούν προηγούμενη ασφάλιση προκειμένου να ε, δεχθούν την ταξινόμηση ενός οχήματος. Ο Πρόεδρος. Ωραία. Δεν θα ξεκινήσουμε τώρα δεύτερο γύρο ερωτήσεων ε, προς την ε, Κομισιόν. Λοιπόν, ο κύριος Λούις, ε, ορθώς ε, εάν παρατηρήσει κανείς ε, τις ε, μετακινήσεις των οχημάτων ορθώς διαπιστώνεται ότι τελικά υφίσταται κυρώσεις ας πούμε η χώρα ταξινόμησης. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να απαντήσουμε στα προβλήματα της ζήτησης χωρίς υπερβολικές χρεώσεις. Όσον αφορά την απώλεια εσόδων στην ουσία θα δημιουργηθεί νέο έσοδο ε, γιατί ε, ε, θα μετακινείται η ταξινόμηση εντός των συνόρων όσον αφορά το leasing θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να αγοράσει αυτοκίνητο σε μια χώρα να το πουλήσει σε μια άλλη και επομένως δημιουργείται μια νέα αγορά η οποία θα δημιουργήσει προσθέμενη αξία. Ε, δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει από την ομάδα του Brainport. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα είναι γεγονός ότι ε, έχοντας πιο πιο καλό ας πούμε φωτογραφικό υλικό μπορεί κανείς ε, να έχει καλύτερες κάμερες. Από την άλλη πλευρά η προστασία των ε, προσωπικών στοιχείων βεβαίως είναι κάτι που η κάθε χώρα θα το αποφασίσει. Όσον αφορά την ιδιωτική εταιρική σχέση πρέπει να σας πω ότι ε, ας πούμε όσον αφορά την ασφαλή λωρίδα, δηλαδή την, τη δεξιά λωρίδα έχουμε μεγάλη μείωση της χρήσης της λωρίδας αυτής και νομίζω ότι αυτό είναι ε, σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Ευχαριστούμε τους ομιλητές της ε, πρώτης, ε, του πρώτου τμήματος της ακροασίας μας. Εάν έχουμε χρόνο, ενδεχομένως θα μπορέσετε να απαντήσετε, να έχουμε και άλλη συζήτηση. Τώρα, θα μπούμε σε πιο εξειδικευμένα στοιχεία όσον αφορά την ίδια την επαναταξινόμηση. Έχουμε μαζί μας τον Γιώχαν ε, Χάχενμπεργκ, ο οποίος ε, είναι γενικός ε, μάνατζερ της αρχής η οποία ασχολείται με τις οδικές μεταφορές των κάτω χωρών. Ε, ε, χρησιμοποιούνται οι πινακίδες για ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών και υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά ε, και τα οποία σχετίζονται ας πούμε με τις κλοπές αυτοκινήτων κλπ. Έχουμε επίσης μαζί μας τον Ken Fekhoizen ο οποίος ασχολείται περίπου με τα ίδια πράγματα από την πλευρά του Βελγίου όμως. Λοιπόν, θα μιλήσουν οι δύο ομιλητές μας, θα έχουμε ερωτήσεις, απαντήσεις και μετά το κλείσιμο το συνολικό. Πρώτα απ' όλα λοιπόν στο, δίνω το λόγο στον κύριο Γιώχαν Χάκενμπεργκ. Χωρίς μικρόφωνο κύριος Χάκενμπεργκ. Ναι, είμαι General Manager της RDV. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ε, ε, πρόσκληση την οποία μου απίφθηνε αρχικός ο κύριος Τόιν Μάντερς αλλά βεβαίως και ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι σαν δημόσια αρχή για την ταξινόμηση των οχημάτων και των ασφαλιών καθώς επίσης και των αδειών οδήγησης. Ε, αλλά ασχολούμαστε και με την εποπτεία των δρόμων και τους ελέγχους. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά λοιπόν το θέμα. Αυτή τη στιγμή θα εστιάσουμε ε, στην, στο θέμα της μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων ε, ταξινομημένων σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η Ευρωπαϊκή ε, Οργάνωση ε, για το εμπόριο των αυτοκινήτων ασχολείται από κοντά με το θέμα αυτό. Ε, στα αυτοκίνητα τα οποία πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 25% προέρχεται από κάποια άλλη χώρα, κυρίως δε από ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παραμείνει σαφές το σύστημα ταξινόμησης, να καταπολεμηθεί η απάτη και να συμβάλλουμε με τα νέα συστήματα σε καλύτερη οδική ασφάλεια χαμηλό κόστος, ε, υψηλό ε, επίπεδο προσφοράων υπηρεσιών προς τους ε, πολίτες μας. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και πιστεύουμε ότι αυτή η νέα οδηγία μπορεί να μας, επιτύχει, μπορεί να μας βοηθήσει συγγνώμη, να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Επομένως καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Κομισιόν. Είναι σημαντικό η ταξινόμηση σε άλλες ενουσιακές ε, χώρες ε, να απλουστευτεί όχι για μας μόνο που είμαστε η αρχή ταξινόμησης αλλά και για τους πολίτες οι οποίοι όλο και περισσότερο ταξιδεύουν εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, θέλει να αγοράζει αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται, να γίνει δηλαδή πιο, πιο απλή η διαδικασία, να απλουστευτούν οι διαδικασίες αυτές και ε, να μπορέσει η μια χώρα να βοηθήσει την άλλη. Η ε, απλούστευση, η απλοποίηση της μεταφοράς ε, οχημάτων από τη μία χώρα στην άλλη έχει ήδη ξεκινήσει και βεβαίως βασίζεται και στην ψηφιακή μεταφορά δεδομένων. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε σήμερα για αυτήν την ανταλλαγή ε, στοιχείων. Εδώ και 20 χρόνια ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τα οχήματα στα πλαίσια των κλεμμένων αυτοκινήτων, των προστήμων ε, και ε, ε βεβαίως όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ και ανταλλαγές μεταξύ των χωρών η αρχή οδικών μεταφορών της Ολλανδίας την οποία εκπροσωπώ ασχολείται με την εξέβρεση ενός συστήματος που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα πλαίσια ε, των, ε, των προνοιών της οδηγίας. Για να καταλάβετε καλύτερα θα σας δείξω ένα σύντομο φιλμάκι.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 Υπάρχει και κάτι το οποίο δεν το είδαμε στο φιλμάκι. Το σύστημα Ιουκάρις ε, συμπεριλαμβάνει και στοιχεία ε, για την ε, ασφάλεια των οχημάτων. Συζητήθηκε το θέμα αυτό προηγουμένως. Όπως είδατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί το γιουκάρι σε συνδυασμό με την οδηγία. Το γιουκάρι χρησιμοποιείται, είναι εύκολο στη χρήση του και έχει αποδείξει ότι είναι ε, ένα καλό σύστημα. Όμως ε, δεν αναφέρεται στη νέα οδηγία της ε, Επιτροπής. Αναφέρεται η οδηγία σε κάποια νέα λογισμικά. Αλλά γιατί να αναπτυχθούν νέα λογισμικά όταν υπάρχουν ήδη αυτά τα οποία λειτουργούν καλά. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι καλό μόνο για την Ολλανδία αλλά και για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η χρήση των υφισταμένων υποδομών και των υφισταμένων δυνατοτήτων πιστεύω ότι μπορεί να σημάνει σημαντική μείωση του κόστους. Το Ιουκάρις έχει στηριχτεί από τα κράτη-μέλη η γνώση της τεχνολογίας, ε, η ευελιξία αλλαγής ε, του ε, λογισμικού, η δυνατότητα εμπλουτισμού των λειτουργιών είναι κάτι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι πρέπει να αναφερθεί το Γιουκάρης στο παράρτημα της οδηγίας. Κάθε χώρα επίσης έχει, συγγνώμη, κάθε όχημα έχει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης ε, πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να ε, περιλαμβάνονται μονάχα απλά τεχνικά στοιχεία, αλλά και να, ε, κατά κάποιο τρόπο να περιγράψετε το DNA του αυτοκινήτου, όλα τα στοιχεία τα οποία θα επιτρέπουν εισαγωγή ή εξαγωγή. Τέλος, στις κάτω χώρες εκτιμάται ότι η απάτη ε, ε, ζημιώνει τη χώρα κατά 150 ε, εκατομμύρια και επομένως πολλά μπορούμε να κερδίσουμε ελέγχοντας τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των αυτοκινητών. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε και για το φιλμάκι. Μάλλον κρύο έκανε όταν γυρίσατε αυτό το φιλμάκι και εκεί ήταν ο πρόεδρός σας που είχε παγώσει. Τι να κάνω. Τώρα. Θα ακούσουμε τώρα κάποιον ε, ειδικό, από το Βέλγιο, που είναι ειδικό λοιπόν στα, στην κλιματικότητα και με τα αυτοκίνητα. Κύριο θα λάβει τώρα το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο... Θέλω, απλώς θέλουμε να, να απλουστεύσουμε τα πράγματα. Ναι, ε, δεν έχει πρόβλημα η αστυνομία, αλλά χρειάζονται. Χρειάζεται η απλοποίηση να μην βοηθήσει του ε, κλέφτε. Εκπροσωπώ την ε, αστυνομία αλλά επίσης και το δίκτυο Κάρπολ που ιδρύθηκε η δυνάμη της απόφασης του Συμβουλίου και εκεί έχουμε ε, μπροχόμενος από όλα τα κρατημέλη Κάναμε επομένως αυτή την μελέτη το 2010 για το δίκτυο Κάρπολ που αφορά το πώς γίνεται το, πώς τέλος πάντων προωθούνται τα κλεμμένα αυτοκίνητα, προηγούμενο ξέπλυμα, ε, ποια, ποιες είναι οι αδυναμίες ε, των ε, σημείων ελέγχου και των, των Υπουργείων Συγκοινωνιών που καταξιώνουν τα οχήματα. Έχουμε ακόμη 653.827 οχήματα τα οποία κλάψουν το 2011. Τα μισά δεν έχουν βρεθεί. Επομένως ακόμα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε επίσης κάποιες επαγγελματικές ομάδες που είναι οι βασικοί εμπλεκόμενοι. Ε, θα πρέπει επομένως να δούμε αυτούς τους επαγγελματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν ε, τεχνολογία ε, και έτσι με ευφύς τρόπους να μπορούν να ξεπλύνουν, να μπορούν να ανακυκλώσουν το συμπίν τα, τα κλεμμένα αυτοκίνητα μέσα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, έχουμε τώρα σημεία ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουν γίνει αρκετά. Ε, όμως το πρόβλημα είναι ότι ε, τα όσα προβλέπονται δεν έχουν υλοποιηθεί. Επομένως, έχουμε το άρθρο 102α του Σέγγεν που ε, που θεσπίζει το, το σύστημα πληροφορία του Σέγγεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αλλά αυτό ε, ε, έχει εφαρμοστεί μόνο από 19 από 25 κρατημέλη και μόνο 9 ελέγχουν το αποδεικτικό της ταξινόμησης και μόνο 11 συστηματικά. Οπότε ξεφεύγουν πάρα πολλά κλεμμένα. Τα είπαμε για το Γιουκάρες, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, αλλά μόνο 14 κρατημέλη μετέρχονται αυτή τη λύση, το Γιουκάρες. Τεχνική έλεγχη δηλαδή, οι οποίοι ε, γίνονται όσον αφορά την επαναταξινόμηση. Αυτό είναι καλό. Όμω η πλαστογράφηση γίνεται πάρα πολύ καλά. Αυτοί που τα κάνουν ε, βρίσκονται σε πάρα πολύ ψηλό. Θα πρέπει κανεί να είναι πραγματικά εμπειρογνώμων. Σε κάποιε χώρε έχουμε ιδιωτικέ εταιρείε που προσλαμβάνονται, όπω στη Σλοβενία, για να ελέγξουν αυτά τα, τα έγγραφα. Αλλιώ ο μέσο υπάλληλο και ο αστυνομικό δεν μπορεί να τσεκάρει το κατά πόσον έχουμε πλαστογράφηση εγγράφων κλείμενο αυτοκινήτου. Τώρα για να δούμε ε, ποια είναι η μέθοδος ξεπλήματο και γιατί μπορούμε να κάνουμε πρώτα πρώτα. Εάν δεν έχουμε στο γραφείο ταξινόμησης ε, κάποιο έλεγχο με το SIS ή με το UCARIS ε, κάποιο κλείμενο αυτοκίνητο μπορεί να το ταξινομήσει. Επομένω θα πρέπει να γίνει κάποια έλεγχη. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα εν μέρη θα πρέπει επομένω να χρησιμοποιηθεί το σύστημα UCARIS το SIS. Πρώτον. Δεύτερον, ε, κάποιος πάει και, και φτιάχνει ε, φτιάχνει ένα, για ένα κλεμμένο αυτοκίνητο φτιάχνει ένα πλωστό, ένα φανταστικό, φτιαχτό ε, έγγραφο. Αλλά κάποιος τσεκάρει μέσα το γιουκάρις και διαπιστώνει ότι αυτό δεν, δεν υπάρχει το αυτοκίνητο το οποίο περιγράφεται στο φτιαχτό έγγραφο. Να λοιπόν πώς γίνεται. Και έχουμε επίσης και κάποια έγγραφα ταξινόμηση κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε, το Ιουκάρις αντιμετωπίζει αυτές τις μεθόδους ανακύκλωσης. Γίνεται διασταύρωση επίσης με το κράτος προέλευσης και κανείς αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κάτι στραβό. Τώρα, κλωνοποιημένο χυμβός λέγονται. κάποιος παίρνει τα στοιχεία από κάποιο έγγραφο και τα μεταφέρει σε κάποιο που μοιάζει πάρα πολύ. Έτσι ανακυκλώνεται επομένω το, το όχημα. Γιατί κάποιο του έχει βάλει τα στοιχεία κάποιου μη κλεμμένου οχήματο. Οπότε έτσι βλέπουμε ε, το ότι χρειάζεται να υπάρχει σημαντικό έλεγχο και συνεχώ. Τώρα, επίση, άλλο άλλος τρόπο. Δεν κλέβονται τα έγγραφα. Γιατί κανείς αγοράζει ένα κατεστραμμένο αποτύχημα αυτοκίνητο και στο κλεμμένο του δίνει τα στοιχεία του κατεστραμμένου. Και κανείς έτσι πάει σε κάποια χώρα, το, το ταξινομεί, κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ε, δεν έχει τυπήσει κανένα καμπανάκι ε, σε σχέση με την κλοπή. Θα πρέπει όμως κανείς μέσω του γιουκάρης να μπορεί να ελέγξει το καθεστώς που διέπει το αυτοκίνητο. Επομένω, αν εμφανιστεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο και εμφανιστεί ω ε, ελαφρώ μεταχειρισμένο, τότε χτυπάει το καμπανάκι ότι κάτι στραβό πάει το αυτοκίνητο. Τώρα, επίση, η απάντηση σχετική με τη χρηματοδοτική μέσταση το έχουμε συζητήσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα πάρα πολύ απλό κόλπο. Έχει κανείς ένα συμβόλαιο λίγων μηνών για τέτοια μίσθωση leasing. Πάει κανείς, ταξινομεί το αυτοκίνητο κάπου αλλού. Το αυτοκίνητο φυσικά δεν είναι κλεμμένο, οπότε αν κανείς το ταξινομήσει αλλού και κανείς έχει ένα πλαστό ε, έγγραφο πώλησης, τότε μπορεί να το αλλού πολλές φορές. Του δίνουν και κάποιο είδου προσωρινές πινακίδες, ε, πολύ συχνά γερμανικές πινακίδες και ξεκινάει κανείς την ταξινόμηση ισχυριζόμενος ότι είναι ε, αυτοκίνητο που έχει κάποια εταιρεία. Όμως μετά από κάποιους μήνες η εταιρεία του leasing θα καταγγείλει την εξαφάνιση του αυτοκινήτου, αλλά έχουν περάσει κάποιοι μήνε και έχει διταξικονομηθεί το αυτοκίνητο. Το ίδιο εδώ χρησιμεύει για την πόλη. Κανείς μπορεί να δει ότι ε, το εκεί που έχουμε την πινακίδα την προσωρινή, πριν υπήρχε κάποια ας πούμε ιταλική πινακίδα. Και ότι είναι αυτοκίνητο το οποίο έχει ε, χρηματοδοτική μίσθωση στην Ιταλία πριν την πινακίδα. Και έτσι με το u μπορεί κανεί να δει αν έχει κλαπεί ή όχι, αν είναι κατεστραμμένο το αυτοκίνητο ή αν έχει κλαπεί το έγγραφο ταξινόμησης επί του παρόντο. Αυτά προβλέπονται στο παράρτημα του σχεδίου της πρότασης κανονισμού. Και κατά αυτόν τον τρόπο ε, μπορούμε να πούμε ότι έτσι έχουμε το πρώτο υποχρεωτικό έγγραφο είναι κάτι πέρα από το UCARIS ή το SIS και έτσι θα έχουμε επομένως υποχρεωτικούς συστηματικούς ελέγχους. Και έτσι θα κάνουμε πάρα πολύ δύσκολο να ανακυκλωθεί το αυτοκίνητο, να ξεπληθεί και έτσι θα χτυπήσουμε ε, τα κυκλώματα αυτά των εγκλήματος. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας μιλήσω σε σχέση με το ποια σκοτεινή πλευρά της ελεύθερης αγοράς. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ πρακτικά όσο μα είπε ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις πληροφορίες. Από την πρώτη γραμμή θα έλεγα του πυρός. Και περιμένω να ακούσω και τους συναδέλφους και τις θέσεις σας. Έχουμε χρόνο λοιπόν τώρα στη διάθεσή μας. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Ο κύριος Μάντερς. Μετά η Κάθριν, ο Ανδρέας. Ο κύριος Σόβερ είναι και αυτός εδώ. Κύριε Μάντερς, πρόεδρε ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον το πώς ε, προχωρεί μέσα στην έκθεση αυτή η τεχνολογία. Δύο ερωτήσεις. Μία γενική καταρχάς. Είναι δυνατόν αυτή η ευφυής κάμερα που έχετε συνδεδεμένη στο σε παραδείγματι, αλλά φαντάζομαι ότι ελέγχεται από τον υπολογιστή η πινακίδα, έτσι δεν είναι, όχι από κάποιον υπάλληλο που κάθεται μπροστά σε μια οθόνη. Αυτόματο υπολογιστή ε, διασταυρώνει με τα στοιχεία που έχει μέσα στο σύστημα του YouCares για να βελτιστοποιείται ο έλεγχος. Αυτή είναι η ερώτησή μου η πρώτη. Και δεύτερον, μιλάμε για προσωρινή ταξινόμηση και ρωτώ εάν είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ψηφιακή ταξινόμηση ώστε να μην τα χρειαζόμαστε. Αγοράζει δηλαδή κάποιο ένα αυτοκίνητο, γίνεται ταξινόμηση. Και εδώ νομίζω ότι δίδεται απάντηση και στην ερώτηση της Κάθριν. Το κράτος μέλος όταν έχει την ταξινόμηση ψηφιακή αυτόματα ζητεί και την καταβολή του σχετικού τέλους. Δεν υπάρχει δηλαδή προσωρινή ταξινόμηση, δηλαδή ξεφεύγουμε από αυτή, το, αυτή την κρίζα ζώνη χάρη στην τεχνολογία, την κρίζα ζώνη της ε, προσωρινής ταξινόμησης. Και αυτό πάλι ήταν ερώτηση. Και για τους έξι μήνες που έχετε ήδη καταβάλει, λέει ο Πρόεδρος. Μάλλον δεν έχουν συστήματα επιστροφής χρημάτων τα, οι δημόσιες αρχές μόνο για συλλογή. Ο κύριος Σφάπ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο που μας παρουσίασε αυτή την ωραία ταινία εδώ. Μέχρι στιγμής στο Ιούκαρις ε, συμμετέχουν όλα τα κρατη Μάλλον όχι από ό,τι κατάλαβα. Α, θα μου πείτε αν είναι σωστό εάν συμμετέχουν όλα τα κρατη όχι και γιατί δεν συμμετέχουν όλα. Ο πρόεδρος, νομίζω το είδαμε ήδη από το βίντεο, αλλά η γενικότερη ερώτηση, και φαντάζομαι την ε, περιμένε ο εισηγητής, ο ομιλητής, και που δεν περιλαμβάνεται στην ε, πρόταση, αλλά ασφαλώς ενδιαφέρει. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια βάση μόνιμη δεδομένων. Η κυρία Στάιλερ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους δύο ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Είπατε 14 κράτη-μέλη και εγώ όπως ο κύριος Φαπ θα ρωτήσω εάν δεν ανήκουν όλα τα κράτη-μέλη γιατί είναι αυτά που δεν ανήκουν στο Σέγγεν ενδεχομένως. Οι συμμετέχουν ενδεχομένω κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ισλανδία, Φερρυπίν. Συνεργάζονται και αυτά. Μας είπατε ότι τα μισά από τα αυτοκίνητα που ανακτώνται έχουν κλαπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς πρέπει να δούμε αυτό πιο λεπτομερώς. Τα κράτη-μέρη δηλαδή τον τα οποία ε, σημειώνουν μεγαλύτερες κλοπές από ό,τι κάποια άλλα. Μπορείτε να μας τα πείτε και ίσως αν υπάρχει κάποια εξήγηση ή υπάρχουν κάποιες βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα αποτροπής ή εν πάση περιπτώσει πώς μπορούμε να έχουμε ενημέρωση για το ποιες είναι οι συμμορίες που δραστηριοποιούνται στην κλοπή οχημάτων, τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ λοιπόν για την πληροφορία. Είναι δυνατή. Βέβαια πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ζητήματα τα οποία προκύπτουν αναγκαστικά στη χρήση του συστήματος αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε πάντως, ε, κυρία Ρίλε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, την πολύ καλή, τις πολύ καλές παρουσιάσεις που αποτελούν και μια πολύ καλή βάση για να αρχίσουμε την εντατικότερη ε, ενασχόληση με το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σόμπερμαϊρ, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω και εγώ και θα ήθελα να πω ότι στην ε, έναρξη της ταινία υπήρξαν κάποια σημεία τα οποία δεν μου έδωσαν αρκετές πληροφορίες. Θα ήθελα λοιπόν πιο πολλά στοιχεία για το ποιος είναι σε ποιον ανήκει το σύστημα, ποιος διαχειρίζεται το σύστημα και σε ποιο πεδίο κινούμεθα ακριβώς, γιατί μου φαίνεται σαν μια λογική, πρόσθετη βέβαια, ε, λύση. Επίσης με ενδιαφέρει και θεώρησα πολύ ενημερωτική την παρουσίαση από τον ε, κύριο της Ολλανδικής Αστυνομίας που παρουσίασε διάφορα ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν αυτές οι πληροφορίες που μας δώσατε με τους πίνακες σας μπορούν να διατεθούν και σε πιο αναλυτική μορφή για να έχουμε πιο πολλά στοιχεία γιατί θα ήθελα να ρίξουμε φως αυτά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγετε, τι ακριβώς χρειάζεται, τι είδους προτάσεις ή ενδεχομένως υποδείξεις θα μπορούσατε να προσφέρετε. Αυτό θα με ενδιαφέρε ως ε, συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με την πρότασή σας. Ο Πρόεδρος. Σκοπεύω και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Εσείς είστε σκιώδης βεβαίως. Ναι, αν ε, σκεφτόμουν το Γιωκάρης ε, αν μπορείτε να μου πείτε, ναι, ακριβώς ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του Γιουκάρης. Το Γιουκάρης μπορεί να είναι, ας πούμε, ευρωπαϊκός οργανισμός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Αν μπορούμε να βάλουμε την ιδέα αυτή ε, και στον κανονισμό, καλό θα ήταν να ξέρουμε ε, τι γίνεται, γιατί έχουμε και τους κανόνες του ανταγωνισμού κτλ. Δηλαδή ε, η Κομισιόν, ε, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον θα ήταν ε, οι ιδιοκτήτες του Ιουκάρης. Ναι, αλλά παραμένει το πρόβλημα ότι μπορεί τα κράτη-μέλη να θέλουν έναν άλλο τρόπο ας πούμε, λειτουργίας που θα είναι δικός τους. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Να επανέλθω στον κύριο Βακχάουζεν. αναφέρθηκε σε κάποιες... Ε, ο κ. Βακχόιζαν αναφέρθηκε ε, σε απάτες και είπαμε ότι θα πρέπει τα στοιχεία του αυτοκινήτου λέμε να μπαίνουν στο παρμπίζο του αυτοκινήτου να μπορεί να τα δει ε, η αστυνομία να μπορούν να καταγραφούν τα στοιχεία εύκολα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τεχνολογική, ηλεκτρονική τεχνολογία ε, για την ε, ταυτοποίηση που μπορεί να κρυφτεί ε, εύκολα στο αυτοκίνητο και που μπορεί να την χειριστεί κανείς πάρα πολύ εύκολα. Είναι ένα ζήτημα και αυτό προς συζήτηση. Ωραία, θέλει κανείς άλλος να συζητήσει, να πει κάτι Ίσως ε, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Χάκεμπερκ, ε, όχι μάλλον από τον κύριο Βακχόισεν πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα για τις περισσότερες λεπτομέρειες, πρέπει να πω ότι έκανα μία έκθεση το 2010, ε, την οποία εδώ συνόψισα την έχω επικαιροποιήσει με νέα στοιχεία και επομένως μπορώ ωραιότατα να τη στείλω στην Επιτροπή σας έτσι ώστε να την αναγνώσετε και να δείτε τις περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, εντάξει, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω και κάποια στοιχεία τα οποία ε, είναι έτσι πιο απόρριτα και αφορούν μόνο την αστυνομία. Ε, θα κάνω λοιπόν αυτήν αυτό το ξεκαθάρισμα και θα σας το στείλω. Όσον αφορά την απάτη, ναι, ε, οτιδήποτε, ε, οποιαδήποτε αλλαγή στο σασί ας πούμε θα πρέπει να γίνει με φυσικό ε, τρόπο. Τώρα η βινιέτα η οποία θα είναι ορατή απ' έξω δεν έχει πάρα πολύ σημασία για μας. Δηλαδή με έναν καλό εκτυπωτή μπορεί κανείς να αλλάξει τα στοιχεία αυτά χωρίς κανένα πρόβλημα. Ε, η RFID έχει ε, ιδέες ε, τα τελευταία χρόνια, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν γίνεται πάρα πολύ συζήτηση Ε, η μόνη ευρωπαϊκή ιδέα ήταν ε, να πασπαλιστεί το αυτοκίνητο με διάφορα σωματίδια ε, τα οποία υπό ειδικό φως θα μπορούσαν να φαίνονται. Αλλά ήταν διστακτικός ο τομέας όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του προγράμματος ας πούμε. Αυτή τη στιγμή γίνονται μελέτες. Ξέρουμε ότι και η Κομισιόν ε, ήθελε να κάνει κάποια σχετική μελέτη αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έχουμε νέα για το κατά πόσον προχώρησε. Επιτροπή ε, αυτό απαντά στην ερώτησή σας για το RFID. Κύριε Χάκενμπεργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τον αριθμό των κρατών μελών ζητήσατε να μάθετε που συμμετέχουν στο Ιουκάρις. Είναι 14. Έχουμε άλλωστε και τη συνθήκη Πρύμ που μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ε, το Ιουκάρις ε, και εκεί στην με αναφέρεται ότι ε, υπάρχει υποχρέωση χρήσης του γιουκάρις. Αυτή τη στιγμή έχουμε 19 χώρες μάλλον που συμμετέχουν στο Ιουκάρις. Και έχουμε και άλλες 6 χώρες οι οποίες θέλουν να συντονιστούν με το σύστημα Ιουκάρης. Αυτός ο συντονισμός θα γίνει φέτος κάποια στιγμή και έχουμε και δύο χώρες, και δύο χώρες αυτές που ε, λείπουν από τις 27 δεν αποφάσισαν ακόμα να χρησιμοποιήσουν το Ιουκάρης. Αλλά θα πρέπει να το κάνουν υλοποιώντα τη συνθήκη πρίμ Η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι αυτές οι δύο χώρες. Αυτά όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, ποιο, δεύτερη ερώτηση. Ποιος είναι ο χρηματοδότης, ο ιδιοκτήτης. Υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει μάλλον... Ναι, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των ε, ε, κρατών μελών και των ιδιοκτητών ε, και από κοινού αποφασίζουν ε, μέσω μιας διοικητικής επιτροπής ε, για τα νέα στοιχεία τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα. Ε, δεν είναι ακριβή η συμμετοχή, είναι περίπου 100.000, κάτω από 100.000 για κάθε χώρα μέλος. Ξέχασα να πω ότι σύμφωνα με τη συνθήκη πριν ήδη πληρώνει εισφορά η κάθε χώρα και επομένως με τον τρόπο αυτό βοηθούνται όλοι να μείνουν συνδεδεμένοι στο σύστημα. 30.000 ε, ε, στην ουσία κοστίζει η συμμετοχή των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη είναι οι ιδιοκτήτες, αυτοί αποφασίζουν ε, τις νέες εξελίξεις, αυτοί αποφασίζουν τις λειτουργίες που θα έχει το σύστημα κτλ. Τελευταία ερώτηση σχετικά με την διασύνδεση με τις αυτόματες κάμερες Αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει κάποια δυνατότητα διασύνδεσης, δεν ξέρω αν γίνεται σε πραγματικό χρόνο real time. Ο γείτονά μου εδώ μπορεί, που είναι ειδικό για κάμερες ίσως μπορεί να σας πει μερικά πράγματα περισσότερα. Και επίσης υπάρχει η δυνατότητα από όσο, ε, γνωρίζουμε αυτόματης λήψης των ε, φωτογραφιών χωρίς μεσολάβηση ανθρώπου. αυτά. Σχετικά με το Ιουκάρις πάντα. Υπάρχει ας πούμε κάποια κεντρική υπηρεσία, υπάρχει κάποια κεντρική δομή. Όχι, δεν είναι κεντρικοποιημένο σύστημα. Έχουμε την Participants Board ε, που είναι κατά κάποιο τρόπο μια κεντρική επιτροπή χωρίς να είναι όμως στην ουσία ε, κεντρική επιτροπή. Ε, χρησιμοποιείται το δίκτυο Testanet για να, για να μεταφέρονται τα στοιχεία από τη μία χώρα στην άλλη και υπάρχουν και διάφορα ε, λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούμε που προέρχονται είτε από τη συνθήκη ΠΡΟΥΜ είτε από τον ε, κατάλογο ε, αδειών οδήγησης Ε, ο καθένας στο δικό του υπολογιστή έχει σύνδεση με το δίκτυο και έχει ε, και ε, διασύνδεση με την Κεντρική Τράπεζα Δεδομένων, με τα στοιχεία ταξινόμησης. Είναι πολύ απλό το λογισμικό. Και στην ουσία αποτελεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο. Θέλετε να πείτε κάτι, ναι. Οι 14 που ανέφερα ήταν τα κράτη-μέλη της συνθήκης για πληροφορίες και ανταλλαγή. Δηλαδή είναι μόνο των ε, ε, υπηρεσιών ε, επιβολής του νόμου. Δεν υπάρχει υποχρέωση όμως για μια υπηρεσία ταξινόμησης να επαληθεύει. 14 λοιπόν είναι οι χώρες, οι οποίες η αστυνομία έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Μετά πάμε στις 17, 27, που βεβαίως εάν και 27 έχουν το Ιούκαρις θα, είναι, θα έχουμε λύσει λίγο πολύ τα προβλήματα. Μια φράση να σας πω, από ό,τι γνωρίζω, δεν χρειάζεται να προσχωρήσει κανεί στην, στην συνθήκη για να χρησιμοποιήσει το Ιούκαρις. Είναι καλά και καθόλου διαφορετικό. Καλά είναι αυτό ένα θέμα. Και, ο, ο κύριος Επιτροπή θα μας το διευκρινίσει. Κύριε Φαντελά. Ναι, για να επανέλθουμε στην αυτόματη αναγνώριση των πινακίδων. Αν δεν τι γίνεται σήμερα, όσον αφορά την έλεγχο του ορίου ταχύτητος, αυτό γίνεται περισσότερο ε, από ψηφιακά μηχανήματα παρά από ανθρώπινα μάτια. Επομένως, πρόκειται για κάτι το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια η ψηφιακή αναγνώριση. Δεν, δεν ε, προβλήματα. Και έτσι μπορούμε να δούμε αν έχουμε το, ε, ότι σωστές να γίνει στο σωστό όχημα. Ήδη επομένω υπάρχει η βάση δεδομένων, ήδη γίνεται κάτι τέτοιο σήμερα. Δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό το σημείο. Πρόεδρος. Ναι, τα, τις λεπτομέρειες του οχήματο μπορεί να τις δει γιατί αν έχει κάποιες αλλάξει πιναγίδες θα είναι χρήσιμο να δει κανείς τις λεπτομέρειες του οχήματο και αυτά να είναι σε κάποια βάση δεδομένων. Όποτε υπάρχει υποψία που βαρύνει κάποιο όχημα. Κύριε Λούς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πάρα πολύ ευχαριστώ το ότι έχει γίνει τόση πρόοδος όπως λέει ο αστυνούγας από το Βέλγιο και έχουμε τόσο μεγάλη μείωση στα ε, κλεμμένα αυτοκίνητα. Το θέμα είναι λοιπόν όταν κάποιος έχει νομίμως ε, καταβάλει το, το, για το, για το leasing, αλλά έχει σκοπό μετά να το ιδιοποιηθεί. Εδώ είναι το δύσκολο. Και αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε εδώ είναι το πώς θα, θα βελτιώσουμε τη διαδικασία, ούτω ώστε να έχουμε τεχνικούς τους καλύτερους, πως θα χρησιμοποιούν περισσότερη τεχνολογία για πρόληψη της κλοπής. Επίσης, δεν είναι δυνατόν μέσα με τον κανονισμό βέβαια να προστατεύσει κανείς τις εταιρείες leasing ως αφορά τους κακούς πελάτες. Υπάρχουν οι βάσεις δεδομένων και έτσι μπορεί κανείς να ταυτοποιήσει ε, τους, τους, ε, κακούς πελάτες και να μην τους ξανα ε, τους ξαναεκμισθώσει ε, αυτοκίνητο, αλλά τέλος πάντων πόσο παραπάνω ε, προσέχουμε τις εταιρείες όταν οι ίδιες βάζουν τα κριτήρια για τις αλλαγές τους. Μέι. Πολύ σημαντικό. Για τα ζητήματα σχετικά με την τεχνολογία, αναγνώριση οδηγού, αναγνώριση οχήματος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι βασικές αρχές τις προστασίες των προσωπικών δεδομένων να τηρούνται, να μην παραβιάζονται. Για δε την απάτηση σχέση με τον ταχογράφο είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ και θα ήθελα να επισημάνω ότι μία βάση δεδομένων θα μπορούσε, εφόσον το επιτρέπει η τεχνολογία, να είναι μια πολύ καλή λύση και εμείς βέβαια θα ήμασταν διτεθειμένοι να ειναι μια πολυ καλη λυση και εμεις δεν θα ημασταν διτεθειμενοι να συνεργαστουμε σε αυτήν. Ο Πρόεδρος και ο κύριος Βόκερ. Επιτέλους, για να τον ακούσουμε πριν από τον εισηγητή, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες είναι όλες ε, οι εισηγήσεις που έγιναν. Και για το Γιούκαρις, ίσως πρέπει να πούμε πρώτα-πρώτα ότι όντως η πρόταση όσο έχει σήμερα αφήνει ανοιχτό το θέμα του άρθρου 7 όσον αφορά δηλαδή τις εφαρμοστικές πράξεις κομισιών που θα πρέπει να προτείνει για το τι γίνεται όσον αφορά το software της βάσης δεδομένων για να εφαρμοστεί να υλοποιηθεί ο οργανισμός. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει ακόμα ε, και δεν είναι το θέμα του Ιουκάρης και έχουμε όντως στο παρελθόν την, την, την χρήση σε διαφορετικούς τομείς του Eucharist. Οπότε, γιατί να μην χρησιμοποιηθεί το Eucharist στα πλαίσια ε, αυτού του νομοθετήματος. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της και αυτή την εκδοχή. Να δούμε τι επιλογές έχουμε για ούτως ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να επισυμπιέσουμε τα έξοδα τα σχετικά με την χρήση της βάσης δεδομένων. Τώρα όσον αφορά ε, αυτά τα σχετικά με την προσωρινή ταξινόμηση, αν μπορεί αυτό να εξαλειφθεί, έχουμε τώρα μία μεταβατική λύση. Από πρακτικής πλευράς είναι δύσκολο να κάνουμε αυτό που είπατε γιατί θα σήμαινε αυτό ότι το κράτος μέλος ταξινόμησης θα πρέπει να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό νέο για λογαριασμό του κράτους προορισμού του οχήματο. Οπότε, κατά γνώμη μας, αυτό το προσωρινό ε, έγγραφο υποζωνές πινακίδες χρειάζονται. Όμως τα πράγματα θα διευκολυνθούν με τη βάση δεδομένων. Τώρα αυτό που είπε η κυρία Μέη στον προηγούμενο γύρο ερωταπαντήσεων, ναι, η βάση δεδομένων προβλέπει πληροφορίες για την περίοδο ισχύω του πιστοποιητικού και επίσης όσον αφορά κάποια πιστοποιητικά τα οποία ε, έχουν ανακληθεί. Άρα και αυτό θα κρυφθεί ότι βάση δεδομένων. Ο Πρόεδρος. Να ευχαριστήσουμε όλους τους αγορετές εκτός από εσάς, διότι βοηθήσατε και συμβάλλατε στην ακροασή μας, που είναι πάρα πολύ ωφέλιμη και είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπο να αρχίσει η νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Τώρα την τελευταία λέξη την έχει ο συγητής ο κύριος Μάντες. Και επίσης να δούμε πώς θα πάει το χρονοδιάγραμμα για, το, για την έκθεση που έχει ακόμα προσωρινό χαρακτήρα και θα εγκριθεί οριστικά από τους ε, συντονιστέ. Βεβαίω είναι και το θέμα του χρονοδιαγράμματο του Συμβουλίου. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τι ε, ενεργέ μα. Ο κύριο Μαντέρ. σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλέ πληροφορίε. Θα βρει το φάσμα. Από τη μια θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους πολίτες. Να είναι πιο απλά τα πράγματα και από την άλλη πρέπει να έχουμε και σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις ε, και την υλοποίηση, την επιβολή των όσων αποφασίζονται. Για να συμφωνήσω με την κυρία Ρούλε, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής, όπως έχει αυτή τη στιγμή. Ίσως δεν να ακούσουμε και τους ε, βενζινοπόλες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν μια πρόσβαση βάση δεδομένων για να δούνε αν συμφωνεί ο αριθμός της πινακίδας με τον ε, αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου και αν τυχόν χτυπήσει συναγερμός ότι δεν είναι το, ότι το αυτοκίνητο είναι κλεμμένο να ζητούν πριν από την ε, χρήση της αντλίας στην καταβολή του τιμήματος για τη βενζίνη. Γιατί μερικές φορές είναι και μεγάλα τα ποσά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πληροφορίες, άρθρα, είτε η ΑΝΤΑΚ, είτε η κάθε άλλη αντίστοιχη οργάνωση που υπάρχει στην κάθε χώρα μπορούν να αποτελέσουν καλά μέσα για να καταγράψουμε τα προβλήματα αλλά και να δείξουμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά ε, όσο βελτίωση και να χωράει ήδη λειτουργεί για το χρονοδιάγραμμα. Το έχω συστήσει με τη γραμματεία, δεν το έχω μπροστά μου. Το έχετε εσείς όμως. Ας ε, ορίσουμε λοιπόν τις προθεσμίες, τώρα που δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά, αλλά πάση χρόνο είχαμε, γιατί είχαμε κάποιο θέμα για τις ε, τροπολογίες και τώρα που έχουμε αρκετό χρόνο να διαρχίσουμε σωστικά από την αρχή ας ε, τον αξιοποιήσουμε, ας ε, παραμείνουμε σε επαφή και ας βρούμε λύσεις, προτάσεις. που να είναι αποδεκτές και πρακτικές. Ασφαλώς, αν κάποιε αρχές δεν συμφωνούν, δεν συνεργάζονται δηλαδή, μπορούμε να τις υποχρεώσουμε. Ο πρόεδρος, χρονοδιάγραμμα. Και όπως είπα θα πρέπει να το ολοκλη... να το οριστικοποιήσουμε. Είναι κάπως χαλαρό γιατί, για μένα, αλλά όπως είπατε χρειάζεται χρόνος. Λοιπόν, μέχρι 29 Απριλίου πρέπει να πάει στη μετάφραση η έκθεση. Πολύ χρόνο έχουμε δηλαδή. Έχουμε εξέταση 29-30 Μαΐου, 27 Ιουνίου τις τροπολογίες, 18-19 Σεπτεμβρίου για την εξέταση και την ψηφοφορία τον Οκτώβριο. Να το ξανακοιτάξουμε όμως εγώ αυτό θα έλεγα. Ο κ. μου λέει ότι το Συμβούλιο ενδιαφέρεται πολύ σοβαρά γι' αυτό. Έχει ξεκινήσει σοβαρή δουλειά, εντατική, άρα ίσως μπορούμε κάπως ε, να ε, πιέσουμε. Έχει γίνει τώρα η ακρόαση πλέον, αλλά δεν χρειαζόταν και όλα να γίνει ακρόαση για να έχετε κάποιες ιδέες και προτάσεις. Έτσι λοιπόν μπορούμε νομίζω να προετοιμάσουμε τις θέσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ για όσους έλαβαν μέρος. Ήταν πολλές οι προσπάθειες, πολλοί άνθρωποι ενεπλάκησαν, οργάνωση, οργανώσεις, κάτι μέλη. Πολλοί παρακολουθούν την ακρόαση αυτή και ελπίζω να τη βρήκαν ενδιαφέρουσα και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα ως εκπλήση της προτάσεως. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συνεδρίαση για το πρωί. Θα σας ξαναδώ στις 3 το απόγευμα και ελπίζω να είναι πολύ άριθμοι οι συναδελφοί βουλευτέ. Ο κύριο Σεμέτα, ελπίζουμε ότι θα είναι παρόν. Ξέρουμε ότι ήταν κάπω αδιάθετο σήμερα, αλλά πιστεύουμε να βρει το κουράγιο να έρθει. Παρακαλώ, τρει ακριβώ το απόγευμα να είσαι στην αίθουσα.